Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακαλώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ. Να έχετε υπόψη ότι η απογευματινή μας συνεδρίαση 2 με 5.30 έχει ακυρωθεί. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για την ημερήσια διάταξη, ε, την εγκρίνουμε. Επίσης, ε, διερμηνία. Έχουμε σε όλες τις γλώσσες, εκτός από φιλαδικά, λετωνικά, λιθουανικά και κελτικά. Έγκριση των συστάσεων των συντονισμών. Δυνάμει το άρθρο 214. Η έγκριση των στάσεων των συντονιστών δυνάμει το άρθρο 214. Σας έχουμε στείλει σημείωμα της συνεδρίασης της 21ης Ιανουαρίου του 2020. θα, θα βρείτε το σημείο αυτό στα έγγραφα της συνεδρίασης. Διορισμό ηγητών. Ο Όντρι Κοβάρικ από την ομάδα των φιλελευθέρων Renew Europe ανέλαβε την έκθεση της ΛΥΜΠΕ επί της προτάσεως ε, για απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκορωσίας για τη διευκόλυνση έκδοση θεωρήσεων διαβατηρίου. 219 κάθετος 182. Εφαρμοστικές εκθέσεις. Ο Λοράνς Βίντσε από το ΕΛΚ έχει οριστεί συγητής της γνωμοδότησης της ΛΥΜΠΕ προς επιτροπές ΑΦΕΤ και ΙΝΤΑ για την εντολή των διαπραγματεύσεων σε σχέση με τις μελλοντικές μας σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. 2020 κάθετος 2023. Η Επιτροπή μας εγκρίνει τις συστάσεις των συντονιστών και τις αποφάσεις τους, δυνάμει το άρθρο 214. Ναι, από ό,τι βλέπω. Οπότε περνάμε στο σημείο 3 της σας διάταξης Ερώτηση για γραπτή απάντηση με κωδικό ε00251519 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ερώτηση της κυρίας Κονίλια Έρνστ με θέμα τον Ευρωπαϊκό Έλεγχο της Μετανάστευσης στο Μαρόκο. Αγαπητοί συνάδελφοι, το πρώτο σημείο της ημέρησης διάταξης αφορά μια ερώτηση για γραπτή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα τον Ευρωπαϊκό Έλεγχο της Μετανάστευσης στο Μαρόκο. Την ερώτηση υπέβαλε η κυρία Κονέλια Ένστ από την ΚΟΕ το, στις 2 Αυγούστου 2019 μάλιστα. Παρόλα αυτά δεν ε, ε, λάβαμε γραπτή απάντηση εντός της ε, προθεσμίας των 6 εβδομάδων που προβλέπει η παραγραφος 3 του άρθρου 138. Ελήψη λοιπόν γραπτής απάντησης και δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 138 οι συντονιστές αποφάσισαν να θέσουν το σημείο αυτό στη σημερινή μας ημερήσια διάταξη και να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει προφορικά. Οπότε θα δώσω το λόγο στην κυρία Νταβίνια Γουτ, που είναι τη ματάρχης της Γενικής Διεύθυνσης Home, ε, Διεύθυνση Στρατηγικής και Γενικών Υποθέσεων, Μονάδα Διεθνούς Στρατηγικής. Θα δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο στην κυρία Κονέλια Ένστ που υπέβαλε το ερώτημα για γραπτή απάντηση. Ή μάλλον, ή μάλλον όχι. Πρώτα θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας ε, κύριε Πρόεδρε, εξότιμη Ευρωβουλευτέ. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω ειλικρινέστατα συγγνώμη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθυστέρησή μας ε, στην απάντηση σε αυτό το τόσο λεπτό και το θέμα. Σας διαβεβαιώ ότι η πρόεδρος Φοντερ Λάιεν ζήτησε από όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στην ανάγκη υποβολής γραπτών απαντήσεων στις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Επίσης, η διαδικασία έγκρισης για τη γραπτή αυτή απάντηση ήδη έχει ξεκινήσει και θα δοθεί πολύ σύντομα γραπτή απάντηση στην ερώτησή σας. Αλλά θα μπορούσα ήδη από τώρα να σας δώσω κάποια βασικά στοιχεία. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στήριξε την εθνική στρατηγική του Μαρόκου για τη μετανάστευση και το άσυλο από τη στιγμή που εγκρίθηκε το 2014 με πολλά και διάφορα σχέδια ε, ύψους 342 εκατομμυρίων ευρώ. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν την πρόθεση της προστασίας των μεταναστών και πρόσβαση στη νομική αρρωγή, ενίσχυση της μεταναστευτικής πολιτικής και σε κεντρικό αλλά και σε αποκεντρωμένο τοπικό επίπεδο, η προώθηση του διαλόγου μεταξύ των χωρών του Νότου για τη μετανάστευση, καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης μαζί με την ε, διαχείριση των συνόρων, την καταπολέμηση της λαθροδιακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων. Ε, και το πακέτο 140 ε, εκατομμυρίων που αυξήθηκε κατά 4 εκατομμύρια το 2020 και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δρομολογήθηκε μέσω προγράμματος για τη στήριξη της εφαρμογής της εθνικής ε, μεταναστευτικής πολιτικής του Μαρόκου και στήριξε κυρίως δύο σχέδια. Το ένα ε, υλοποιείται από έναν εθνικό φορέα και μια διεθνή οργάνωση προκειμένου να παρασχεθεί κατάρτιση και εξοπλισμός για τη διαχείριση των συνόρων. Σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό, επικεντρωνόμαστε κυρίως σε οχήματα, ασθενοφόρα και άλλα μέσα μεταφοράς, αλλά και ραδιοεξοπλισμό και ε, δορυφορική ε, ε, δορυφορικό εντοπισμό, καθώς και κάποιο ιατροδικαστικό εξοπλισμό. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με το Μαρόκο και να υλοποιήσουμε πραγματικό διάλογο και εταιρική σχέση σε πολλούς τομείς που αφορούν τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Συνεχίζονται λοιπόν οι συζητήσεις με τις μαροκινές αρχές, προκειμένου να εμβαθύνουμε τη συνεργασία που ήδη έχουμε και την αμοιβαία μας δέσμευση υπέρ της μετανάστευσης, κάτι που αποτελεί πλαίσιο μια ευρύτερη στρατηγική εταιρικής σχέσης. Οι ευρωπαϊκές και Μαροκίνέ αρχές διερευνούν ε, δυνατότητε ανάπτυξη αυτής της συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς Ευρωπαϊκής Ένωση και τους οργανισμούς. Για παράδειγμα, με τον Frontex, την Ευρωπαϊκή Συνοριακή και και την Europol. Γενικώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί να υιοθετήσει μια σφαιρική στρατηγική με τις χώρες εταίρους, συνδυάζοντας όλα τα μέσα πολιτικής, εμπορική, αναπτυξιακή πολιτική, πολιτική θεωρήσεων, ε, συνεργασία για την επανεισδοχή και νόμιμη και προαιρετική ε, μετανάστευση και υλοποίηση και εφαρμογή εταιρικών σχέσεων. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος προς την εκπρόσωπο της Επιτροπής και τώρα να δώσουμε λόγο στην κυρία Έρνστη, η οποία υπέβαλε το αίτημα γραπτής απάντησης και σε άλλους συναδέλφους ε, που τυχόν θέλουν ε, να τοποθετηθούν. Παρακαλώ, επειδή πιέζουμε σε το χρόνο, μην μιλήσετε πάνω από δύο λεπτά. Κυρία Έρνστ, έχετε το λόγο. Δεν θα χρειαστώ καν τα δύο λεπτά, φαντάζομαι. Θα ήθελα να μου πείτε σε τι βαθμό χρησιμοποιούνται και ευρωπαϊκοί πόροι για την ε, ε, οικοδόμηση συνοριακών πραγμάτων ε, και κατά πόσον υπάρχει συνδυασμός των ισπανικών κονδυλίων και ευρωπαϊκών πόρων. Αυτοί οι φράχτες δηλαδή έχουν φτιαχτεί και με ευρωπαϊκά κονδύλια για τις αντισταθμίσεις μάλλον για τις ε, επιδόσεις που περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το Μαρόκο. Έχουμε πετύχει κανένα αποτέλεσμα στις συζητήσεις σε ό,τι αφορά τους Μαροκινούς και το τι θα μας δώσουν ως ε, διαβεβαίωση, τι μέτρα δηλαδή διαβεβαίωσης. Και Ύστερα αυτό που είπατε στην αρχή ότι θα μας ε, στείλετε και γραπτή απάντηση προκειμένου να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για μελλοντικέ χρήσεις. Thank you, Chair. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση να υποβάλω, λέει, κυρία Σπούρεκ, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κάτι που ανακύπτει σε σχέση με το θέμα μας. Το 18 είχαμε 340 παραβιάσεις εις βάρος των μεταναστών από τις αρχές. 79% ε, στα κέντρα υποδοχής. Και έχουμε καταγγελίες ότι το 18 επίσης ε, κρατήθηκαν πάρα πολλοί πρόσφυγες μετανάστες ε, πήραν ε, αποτυπώματα και να τους βάλαν σε λεωφορεία, τους βάλανε χειροπέδες και σε κάποιες περιπτώσεις τους ε, έδασαν τα χέρια με σκηνή και μετά τους εκτόπισαν σε απομακρυσμένες περιοχές και έπρεπε να περπατήσουν ώρες για να φτάσουν στη πρώτη πόλη χωριό. Όμως ε, το Μαρόκο λαμβάνει κοινοτικά κονδύλια από τα ταμεία μας. Δεν ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί το τι γίνεται με τους αλλοδαπούς σε σχέση με το αν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, από πλευρά των Μαροκινών αρχών, ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Θέλει άλλο συνάδελφο το λόγο. Όχι από ό,τι φαίνεται. Οπότε θα ήθελα να σας πω το εξής. Η ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Τροπή από πλευρά της κυρίας Ένστη είναι πάρα πολύ εύστοχη γιατί πρέπει να μας δώσουν κάποιες απαντήσεις και θα μας ήταν πολύ χρήσιμο να μάθουμε πώς αξιοποιούνται τα κονδυλιά μας. Ακριβώς όπως και σε σχέση με την Τουρκία και με τα Βαλκάνια είναι πολύ σημαντική η συνεργασία μας με το Μαρόκο όσον αφορά την πρόληψη για το μεταναστευτικό, όσον αφορά τους ελέγχους και η συνεργασία με τη χώρα αυτά σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές και το πώς θα σταματήσουν αυτές οι ροές προς την Ευρώπη είναι υπόθεση πολύ σημαντική. Άρα θα πρέπει να επενέσουμε τη χώρα για τις προσπάθειες το 18 σταμάτησε το Μαρόκο 74.000 παράμους μετανάστες από το να πάνε στην Ισπανία. Μετά είχαμε επομένω ε, μείωση 60% των ροών προς την Ευρώπη. Επιπροσθέτως, πέρσι 19.500 ήταν οι μετανάστες που διασώθηκαν από το Μαρόκο στην θάλασσα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θέλει να υπάρχει πιο αποφασιστική βοήθεια προς τις χώρες που προσπαθούν να ανασχέσουν την λαθρομετανάστευση. Και είναι επίσης σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι η επανυποδοχή, η, η επαναπροώθηση, η απόθεση τέλο πάντων ε, θα πρέπει να πλαισιωθούν και έτσι να μειωθεί η πίεση των μεταναστευτικών ροών. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε πώς προτεραιότητα τις ε, επιστροφές αυτών των ετούντων άσυλων των οποίων η αίτηση ε, απορρίπτεται. Θα πρέπει να πιέσουμε τις τρίτες χώρες, με τις, ε, να τις πιέσουμε δίνοντάς τους κίνητρα. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάντως θα πρέπει να θέτουμε προϋποθέσεις σε σχέση με τις ε, αποθήσεις, ε, επιστροφές, επαναπατρισμούς. Άρα θα πρέπει έτσι να προσέξουμε τη συνεργασία. Νέα κίνητρα ή ε, αρνητική μόχλευση, αρνητικές πιέσεις. Ευχαριστούμε. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να απαντήσει στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εξιότιμη βουλευτές για αυτές τις σημαντικές ερωτήσεις και επιτρέψτε μου να σας πω κάπως το ιστορικό πλαίσιο των σχέσεών μας με την χώρα όσον αφορά τη μεταστευτική πολιτική. Οι σχέσεις μας ανάγονται στο παρελθόν και υπήρχε μια συμφωνία κινητικότητας το 2013. Οπότε και θεσπίστηκε ένα πλαίσιο συνεργασίας για το θέμα αυτό, για τη μετανάστευση. Και επιβεβαιώθηκαν όλα αυτά σε μια κοινή δήλωση στο τελευταίο Συμβούλιο Σύνδεσης τον Ιούνιο πέρσι. Και η ευρωπαϊκή ενίσχυση προς την χώρα μέσω των προγραμμάτων που ήδη είχαν εκπονηθεί αποτελεί τμήμα αυτού του διαλόγου και εκεί θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι εντάσσεται και η συνεργασία για το μεταναστευτικό καλύπτει όλους τους επιμέρους άξονες της συνεργασίας και την λαθρομετανάστευση και την λαθροδιακίνηση, ε, ε, δουλεμπόριο, προστασία των μεταναστών που ήδη βρίσκονται στη χώρα, ε, καμπάνια για να ξέρει ο κόσμος τι κίνδυνοι υπάρχουν, σωτηρία ανθρωπίνων ζώων που είναι πολύ σημαντικός στόχος για αυτή μας την εταιρική σχέση και ε, αυτό καλύπτει τρίτες χώρες και φυσικά και το Μαρόκο στο δε πλαίσιο της επανεκκίνησης των σχέσεών μας με τη χώρα υπάρχουν κάποια ζητήματα που συζητήθηκαν και περιλαμβάνεται εδώ και αυτό που είπατε πρόεδρε για την επανεισδοχή ε, για τη συνεργασία σχετικά με την επανεισδοχή και υποδοχή εκ νέου αυτών των ανθρώπων και επίσης ε, σχετικές διαυκολύνσεις με τις θεωρήσεις διαβατηρίου και όλα αυτά τα θέματα διαχείριση συνόρων, λαθρομετανάστευση, προστασία, ε, φρενάρισμα του στη, στη λαθροδιακίνηση, δηλαδή δουλεμπόριο, ε, νόμιμη μετανάστευση αλλά και πανυποδοχή, όλα αυτά συζητήθηκαν και οι διάφορες υπηρεσίες ε, τις, που ασχολούνται με την ε, πολιτική ε, δικαιοσύνη και εσωτερικών συμμετέσχουν ε, στις επαφές στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας. Και θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση όσον αφορά την κατασκευή αυτών των φραγμάτων και εμποδίων. Οπότε εμείς πρόκειται, είπαμε και υποσχεθήκαμε και δεσμευθήκαμε να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση για όλα τα ζητήματα της εταιρική σχέσης με τρίτες χώρες. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και αναγνωρίζουμε πλήρως το ότι το Κοινοβούλιο έχει σημαντικό ρόλο πρέπει να ενημερώνεται και πρέπει να απαντήσουμε στο γραπτό σα ερώτημα και σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ κυρία Σίπελ, τώρα το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και συγγνώμη καθυστέρησα λίγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλες τις απαντήσεις που μας έδωσαν τώρα και συμφωνώ απόλυτα ότι η μετανάστευση και το άσυλο είναι ένα πολύ μεγαλύτερο και ευρύτερο κόστο και δεν μπορούμε να το κοιτάξουμε μόνο στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλέ ε, χώρε αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό και υποδέχονται μετανάστε ε, και πρόσφυγε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να το κοιτάξουμε πιο ευρέως το θέμα. Και θα ήθελα να ξέρω τι είδου συνεργασία ε, έχει κατά νου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποια στοιχεία ανέφερε, αλλά δεν μπορούμε να αναφέρουμε, να δεχτούμε μάλλον, ότι ο μοναδικό λόγο για τη συνεργασία σε τελική ανάλυση θα ήταν να αποφύγουμε τι παράνομε μεταναστευτικέ ροέ ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αρκεί αυτό, γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο κόσμο που φεύγει από τα σπίτια του θα πρέπει να έχει μια νέα ευκαιρία για τη ζωή του. Αν θέλουμε να αποφύγουμε λοιπόν την λάθρομετανάστευση θα πρέπει να δώσουμε απάντηση στο πώς μπορούμε να δώσουμε μια νομική απάντηση για αυτούς τους ανθρώπους που διαφεύγουν από τις πατρίδες τους, γιατί στην παρούσα φάση δεν υπάρχει νομιμός τρόπος να μπει κανείς σε μια άλλη χώρα όταν αναγκάζονται να φύγει από τη δικιά του. Και θα θέλαμε λοιπόν να στείλουμε μόνο θετικά μηνύματα, γιατί σήμερα το πρωί και πάλι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων, στη Γερμανία τουλάχιστον, παρουσίασαν και πάλι την προθυμία τους, δήλωσαν την προθυμία τους να υποδεχτούν στις πόλεις τους ε, α, πρόσφυγες ε, από τη Μόρια, για παράδειγμα, και θέλουμε να πούμε ότι θα πρέπει να ε, υπάρχουν όλο και πιο πολλοί οι οποίοι θα συμφωνούν για να γίνεται αποδεκτή αυτή η προσφορά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε την κυρία Ζίπελ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ακράδαντα ότι θα πρέπει να δίνεται ε, καταφύγιο σε αυτούς που ε, διαφεύγουν από εμπόλεμες περιοχές και από ε, καταστάσεις δίωξης. Και με αυτό το γνώμονα δρούμε κιόλα. Και αυτό δεδομένων και των ε, συγκρούσεων και των εμπόλεμων σειράξεων στην ε, γειτονία μας ε, τα τελευταία χρόνια. Να αναφέρω όμω κάτι σε ό,τι αφορά τι ερωτήσει που έγιναν από του βουλευτέ. Να πω ότι έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια νομίμω διαμένοντε Μαροκινού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης και της συνεργασίας αυτής, προσβλέπει στην ανάπτυξη από κοινού με τα κράτη-μέλη στοχευμένων προγραμμάτων για να προωθηθεί η νόμιμη μετανάστευση σε συγκεκριμένους τομείς σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας από τρίτες χώρες και μια σειρά πιλωτικών προγραμμάτων επίσης εφαρμόζονται σε ό,τι αφορά το Μαρόκο συγκεκριμένα. Αυτό λοιπόν αποτελεί μια πτυχή της συνεργασίας η οποία εντάσσεται στην ε, συνεκτική αυτή προσέγγιση, στην ιδέα οικοδόμησης ε, εταιρικών σχέσεων με το Μαράκο και με άλλες χώρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητά άλλο συνάδελφο το λόγο. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης παρουσίαση της έκθεσής μας μετά την αποστολή της Επιτροπής Λίμπες στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογίας των Πληροφοριών μεγάλης κλίμακας στο χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, η Γιουλίσα, στο Τάλιν της Εστονίας, στις 29 30 Οκτωβρίου 2019. Γιατί από την προηγούμενη μας επίσκεψη το 2016 πολλές αλλαγές έγιναν σε ό,τι αφορά τη διαχείριση συστημάτων IT μεγάλης κλίμακας. Και δεν έχουμε μόνο ένα νέο αναθεωρημένο κανονισμό για το eu αλλά έχουμε και πολλά νέα συστήματα που θεσπίστηκαν, ενώ τα παλιά συστήματα αναθεωρήθηκαν ή αναβαθμίστηκαν. Οπότε στο πλαίσιο αυτό η τελευταία μας αποστολή στο Τάλιν, στον οργανισμό Ιουλίσσα, ήταν καλή ευκαιρία για να μας δώσει μια γενική επισκόπηση της εφαρμογής της αναθεωρημένης εντολής και του προγράμματος εργασιών του οργανισμού αυτού, ενώ ταυτόχρονα ενημερωθήκαμε για τα διάφορα συστήματα που διαχειρίζεται ο οργανισμός. Δύο μέλη της ΛΥΜΠΕ έλαβαν μέρος στην επιστολή, η κυρία Σαμπρίνα Πινιεντόλη και ο υποφαινόμενος. Δεδομένου ότι εγώ ήμουν ο επικεφαλής ε, ε, ε, αποστολής και μια και κολλείται η κυρία Πινιεντόλη σήμερα θα κάνω μια παρουσίαση της αποστολής και μετά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους που θέλουν να σχολιάσουν. Καταρχήν, ε, ο κανονισμός 1077 του 2011 ίδρυσε τον ε, οργανισμό αυτό και στόχος του EU είναι να στηρίξει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων με την λειτουργική διαχείριση συστημάτων IT μεγάλης κλίμακας. Το Νοέμβριο του 2018 η εντολή του οργανισμού ενισχύθηκε με ένα νέο κανονισμό τον 2018-1726. Η αποστολή μας στο Ιγιουλίσσα έγινε βάση κανόνων που επιτρέπουν σε τρία μέλη να επισκεφθούν τον οργανισμό στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους ε, στην Επιτροπή και αυτό γίνεται αναδιαιτία και προστίθεται στις κανονικές ποσοστώσεις για αποστολές. Ήταν αυτή η τρίτη μας αποστολή στον οργανισμό μετά την ε, θέση σε εφαρμογή του το Δεκέμβριο του 2012 και η πρώτη ε, αποστολή μας μετά την ενίσχυση της εντολής του στα τέλη του 2018. Η αποστολή μας επικεντρώθηκε στην ε, εφαρμογή του αναθεωρημένου κανονισμού για τον λίσα, στο έργο του Συστήματος Πληροφοριών Σέγγεν 2, στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, το UDAC, το ΕΤΙΑΣ, το ΕΚΡΙΣ. Επίσης, συζητήσαμε και τις μελλοντικές προκλήσεις. Μιλήσαμε επίσης για την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος εργασιών, τις στρατηγικές προτεραιότητες, τη διοίκηση, διακυβέρνηση και τον προϋπολογισμό του οργανισμού Γιουλίσα. Τη δεύτερη μέρα της επίσκεψής μας ε, παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων IT μεγάλης κλίμακας ε, που διαχειρίζεται ο οργανισμός και εστονικές αρχές. Επισκεφτήκαμε το ΣΥΡΕΝ, όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούνται, επισκεφθήκαμε και το αεροδρόμιο του Τάλιν για να εξοικειωθούμε με τη λειτουργία του ΣΥΣ 2, του Σύστημα Πληροφοριών Σέγγεν 2 και του ΒΙΣ στα σύνορα. Ε, ενημερωθήκαμε και για το σύστημα εισόδου-εξόδου της Εσθονίας που λειτουργεί πολύ καλά. Οπότε μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι και τα τρία συστήματα πληροφοριών ε, λειτουργούν καλά και η εισαγωγή νέων συστημάτων επίσης προχωρεί ε, μια χαρά και σίγουρα ο οργανισμός συμβάλλει στην, στην ε, εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων με υψηλό επαγγελματισμό και καλές προδιαγραφές εφαρμόζει το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα θέλαμε να επισημάνουμε τη στρατηγική σημασία που έχει η διαχείριση συστημάτων IT μεγάλης κλίμακας από τον οργανισμό Ιγιολίσα. Επίσης, χαιρετίζουμε την ενισχυμένη σημασία του οργανισμού αυτού που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο άρτιο έργο που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια και στην καλή φήμη που έχει δημιουργήσει. Και επίσης εξετάσαμε κάποια μελλοντικά σχέδια που ίσω ενδιαφέρουν τον οργανισμό. Βέβαια, η αύξηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του οργανισμού θα πρέπει να συνοδευτεί από αύξηση του προσωπικού του και του προπολογισμού του. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυβέρνηση της Εσθονία για την υποστήριξη και τη βοήθεια που πρόσφερε στον οργανισμό και θα την καλούσαμε να συνεχίσει να υποστηρίζει τόσο ενεργά τον Ευχαριστώ και παρακαλώ συνάδελφοι, θέλει κανείς το λόγο για να σχολιάσει. Δεν βλέπω κανέναν. Η κυρία Κέβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η αποστολή της ΕΙΜΠΕ θα έχει την επόμενη εβδομάδα αποστολή στο επιχειρησιακό τμήμα του Στρασβούργου. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε και την αποστολή που κάνατε τον Οκτώβριο στον Ιγιουλίζα στη βασική έδρα, αλλά και στα τεχνικά επιχειρησιακά συστήματα που βρίσκονται στο Στρασβούργο και θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Είναι σημαντικό για να δημιουργήσουμε μια γενική εικόνα των νέων συστημάτων που αναπτύσσονται είτε στον Ιγιουλίσσα είτε στα τεχνικά τμήματα του Στρασβούργου για να εξετάζουμε καλύτερα, ε, καλύτερα την ροή των δεδομένων μέσα από τα σύνορα. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλο συνάδελφο να ζητάει το λόγο. Οπότε, κλείνουμε το σημείο 4 και θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα μέχρι τις 10, γιατί στις 10 θα περάσουμε στη συζήτηση του επόμενου σημείου. Okay, let's start. Ο πρόεδρος. Ας ξεκινήσουμε. Преминаваме към точка 5 от дневния ред. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη παρουσίαση της κατάστασης των πραγμάτων σε σχέση με τη Γενική Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η συζήτηση κοινή και συμμετέχουν ε, οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Δίπλα μου συμπροεδρεύει κύριε Χολμάγερ, όπως γνωρίζετε. Έχουμε τον κονισμό 2017 ε, 39 και αυτό προβλέπει ε, ενισχυμένη συνεργασία και επίσης έτσι ορίζει το άρθρο 18 της Συνδικής για τη Λειτουργία της Ένωσης. Επίσης έχουμε την ε, οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης 2017-1371 και πρόκειται για την μεταφορά ποινικών διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαβέμεις της απάτης στο Εθνικό Δίκαιο. Έχουμε 22 χώρες οι οποίες συμμετέχουν ε, σε αυτό το θεσμικό όργανο. Με μεγάλη μας χαρά υποδεχόμαστε την ε, κυρία Λάουρα Κοντρούτα και έχετε το λόγο κυρία. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε και μου δώσατε την ευκαιρία να έρθω να σας συναντήσω τον Νοέμβριο από τα καθηγοντά μου και το πρώτο που ρώτησα είναι τι πόροι διατίθενται και τι πόροι χρειάζονται ούτω ώστε η Γενική Εισαγγελία να λειτουργήσει τέλη του 2020. Η πρώτη επιστολή που απίφθηνα ε, προς τα κράτη-μέλη ε, είχε ως θέμα το να μου δώσουν κάποια στοιχεία ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι φόρτο εργασία θα έχουμε την πρώτη χρονιά λειτουργία του υπηρεσία μας και οι βασικές παράμετροι που έπρεπε να διαχειριστούμε ήταν ο αριθμός των ε, ε, Ευρωπαίων εισαγγελέων οι οποίοι πρόκειτο να απασχοληθούν στα κράτη-μέλη που συμμετέχουν και επίσης πόσοι θα είναι το προσωπικό της κεντρικής υπηρεσίας στο Λουξεμβούργο. Δεν είναι θέμα τεχνοκρατικό η απόφαση σε σχέση με ε, την χρηματοδότηση. Δεν είναι θέμα ειδικών στα δημοσιονομικά. Πρόκειται να αποφασίσετε για κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πολιτική απόφαση και μην, ε, ε, μην θεωρήσετε ότι είναι κάτι άλλο από το ότι το θέμα είναι οι θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας της υπηρεσίας μας. Και να σας εξηγήσω γιατί γιατί επί τη βάση των στοιχείων που είχα τέλει του περασμένου έτους και σε σχέση με το χρονικό πλαίσιο θα έπρεπε να κάνουμε ε, μια προκαταρτική πρόβλεψη για τις ανάγκες της υπηρεσίας το 20 και το 21. Οπότε εστράφην στην Επιτροπή και ε, τους είπα ότι ακόμα και εάν δεν έχουμε κάποια στοιχεία ε, πάρα πολύ σημαντικά πλευράς κρατών μελών για τη λειτουργία μας, θα πρέπει να αρχίσουμε τη δουλειά. Και αν θέλουμε να ξεκινήσουμε το 2020 θα πρέπει να υπάρξει αύξηση της για αυτή τη χρονιά και θα πρέπει να γίνει ανάλογη προσαρμογή για την πρικοδότηση του 2021. Και σε αυτά τα πλαίσια στις 17 Φεβρουαρίου θα συντηθώ με τον Επίτροπο Reinders. Ήδη ε, έχουμε συναντηθεί επανειλημμένα, ήταν αγαστή η συνεργασία μας και ε, επίσης ε, θα συναντηθώ για πρώτη φορά με τον Επίτροπο Χάν και είναι ξεκάθαρο ότι οι προκατακτικοί υπολογισμοί ε, σημαίνουν ότι το αρχικό χρηματοδοτικό πλαίσιο της συγκρότησης της υπηρεσίας τώρα είναι άχρηστο, είναι κάτι το απαρχαιωμένο γιατί θεωρείται ότι θα ξεκινήσουμε με τους ε, πόρους του 20 και θα λειτουργεί όπως θέλουμε το 23 η υπηρεσία και ότι θα έχουμε χίλιες έρευνες. απαιτήθηκε απαιτήχθη ότι αυτό ήταν εσφαλμένο. Πρώτα-πρώτα, είναι θέμα αρχής. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε μια νομοθετική, κανονιστική υπηρεσία, να αργήσουμε από το μηδέν και σιγά σιγά να εντείνουμε το ρυθμό των εργασιών μας. Πρόκειται περί εισαγγελικής υπηρεσίας θα πρέπει να τηρούμε την αρχή της νομιμότητας, τις ποινικέ δικονομίες των κρατών που συμμετέχουν και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ενεχομένων στις ε, διαδικασίες. Και επίσης θα πρέπει να βελτιώσουμε το επίπεδο προστασίας των χρηματοοικονομικών συμφερών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτω ώστε να υπάρχει ένα σωστό επίπεδο ε, για τις εισαγγελικέ ενέργειες και τις έρευνες σε όλα τα κατημέλη που συμμετέχουν. Και όμως τώρα έχουμε διάφορα προβλήματα σχετικά. Κατά τρίτο λόγο, το ότι τώρα οι εθνικές ένωμες τάξεις ε, πρέπει να καλύψουν και την ε, συγκρότηση της δικής μας υπηρεσίας δεν σημαίνει ότι θα μειωθεί η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, δηλαδή στην πράξη. Γιατί το πρώτο έτος λειτουργίας θα πρέπει να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ε, τη διεκπεριώση 2.000 νέων υποθέσεων και θα κάνουμε έρευνες, θα σκεφτούν ποινικέ διώξεις για κάποιες από αυτές και οι υπόλοιπες θα διαβιβαστούν στις εθνικές εισαγγελικές υπηρεσίες και θα πρέπει από την πρώτη μέρα λειτουργίας να διεκπαιριώσουμε ό,τι είναι της αρμοδιότητός μας και εκρεμεί. Οπότε υπολογίζουμε ότι η υπηρεσία και οι εισαγγελίες της υπηρεσίας μας θα πρέπει να ε, εξετάσουν 3.000 υποθέσεις και να αποφασίσουν σε ποιες θα αναλάβουν ενέργειες και ποιες θα παραπέμψουν. Σύμφωνα με κάποια αυστηρά χρονοδιαγράμματα που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας, επίσης θα πρέπει να μπορέσουμε να συμβάλλουμε με κάποια προσθέμενη αξία, γιατί γι' αυτό συγκροτήθηκε η υπηρεσία μας, αξιότιμοι βουλευτές. Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να τα καταφέρουμε με 32 ε, ε, εισαγγελείς, 22 μάλλον εισαγγελείς και 32 αποσπασμένους εισαγγελείς και 29 άτομα προσωπικό, όπως τώρα προβλέπετε. Για να σας πω συγκεκριμένα τι γίνεται όσον αφορά αυτούς τους αποσπασμένους ε, εισαγγελείς, γιατί είναι κάτι που επανειλημμένα διατυπώνεται και περιέργως διατυπώνεται από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από ό,τι φαίνεται, θα είναι εφικτό, αν όχι προτιμητέο, να δούμε πώς παρά τις δημοσιονομικές ε, δυσκολίες να αρχίσουμε ε, την λειτουργία μας επί τη βάση του τι υποθέσεις ε, διεκπεριώνουν οι εθνικές εισαγγελίες. Σε κάποια κρατημέλη αυτό θα σήμαινε να υπάρχει ένας Ευρωπαίος εισαγγελίας αποσπασμένος που ασχολείται μόνο με αυτό. Μα είναι δυνατόν να, ε, κάποιος να ασχολείται μόνο με κάποιον εισαγγελία που δεν έχει πλήρη απασχόληση σε αυτές τις ε, υποθέσεις που έχει η υπηρεσία μας. Μα τόσα χρόνια που είμαι εισαγγελέα δεν ξέρω αυτό να γίνεται πουθενά στον κόσμο. Δηλαδή να αφιερώνει το εντέρτο της δεστηριοτάς του εισαγγελέα στην υπηρεσία του. Επομένως, ε, κάποιος θα ασχολείται με μία υπόθεση το πρωί, ε, μία ευρωπαϊκή και μία εθνική το απόγευμα και ποιος θα μπορεί να ενεργήσει επιγόντως κάποιες αποφάσεις, ε, ποιος θα αναλαμβάνει την ε, διαδικασία της λειτουργίας ε, όταν είναι στην έδρα του δικαστηρίου. Οπότε, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί στο έργο μας, αν θέλουμε να δώσουμε κάποια προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την πρώτη μέρα λειτουργίας, αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά ανεξάρτητοι, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με κάποιους εισαγγελείς που θα έχουν αποσπαστεί και θα έχουν πλήρη επασχόληση στην υπηρεσία μας, αλλά χρειάζονται τουλάχιστον δύο ένα μέλος. Αυτό ακριβώς καλύπτεται ή προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας μας. Τον Δεκέμβριο μίλησα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και σας ε, ε, ρώτησα αυτό που ρώτησα και τους Υπουργούς Δικαιοσύνης την ίδια μέρα. Τι θέλουμε, να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να λέμε ότι υπάρχει ή θέλουμε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να είναι ένα όργανο αποτελεσματικό. Έχω υπόψη μου ενδιαφέρουσες ε, τροπολογίες που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας επαλλαγής. Νομίζω ότι είναι σωστή κατεύθυνση και ε, αισθάνομαι ε, ότι καλά θα πάνε τα πράγματα γιατί το Κοινοβούλιο θέλει να είμαστε ανεξάρτητοι και αποτελεσματικοί. Ξέρετε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να υπάρχει η υπηρεσία μας και θεωρούν ότι αποτελούμε ένα μέσο εξασφάλισης του κράτους δικαίου στην Ένωση. Μέχρι τώρα διάφορα κράτη-μέλη όσοι συμμετέχουν θέλουν να γίνει αναθεώρηση ε, της πρικοδότησης της ε, υπηρεσίας. Οπότε έτσι θα καταπολεμήσουμε το διασυνορικό έγκλημα, συνεργασία θα έχουμε και περισσότερη εμπιστοσύνη των κρατών μελών, να είμαστε ένα κέντρο αριστείας όσον αφορά ε, επίση τι ε, κατασχέσει προϊόντος ε, εγκλήματος και επίσης την ανάκτηση των οικονομικών ζημιών των κρατών μελών. Επίσης θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα στην καταπολέμηση της απάτης σχετικά με το ΦΠΑ. Και η απάτη αυτή ανάγεται σε 30 με 60 δις ευρώ ετησίως. Νομίζω ότι αξίζει να επενδύσετε στην υπηρεσία μας και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Χολμάιρ τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ συνάδελφε Ράντοφ. Και καταρχάς θα ήθελα να σας ε, καλωσορίσω και να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ζήλο τον οποίο επιδεικνύεται και για τη δουλειά την οποία έχετε κάνει ως τώρα, με την οποία αποδεικνύεται ότι όλες οι προσδοκίες και οι ελπίδες του Κοινοβουλίου που είχαν εναποτεθεί πάνω σας άξιζαν τον κόπο. Θα ήθελα να αναφέρω αυτά που είπατε και εσείς. Εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα έχουμε πολλούς συναδέλφους που επικρίνουν το αρχικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ε, υπονόμευση τάχα του, της Eurojust και της Όλαφ για να τονωθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ξέρετε ότι υπάρχει θέμα υποχρηματοδότησης και ε, υπάρχει υποχρηματοδότηση λοιπόν και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν μπορώ να πω ότι ασπάζομαι αυτή τη λογική. Και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και στην Επιτροπή Κοντ και στην Επιτροπή Προπολογισμού προσπαθήσαμε να συνομιλήσουμε με τους αντίστοιχους ε, επιτρόπους. Ο Επιτρόπος Ότενγκερ μας είχε διαβεβαιώσει ήδη ότι αν υπάρχει ανάγκη σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενδεχομένω να υπήρχε συμπληρωματικό προπολογισμό για την αύξηση των πόρων. Και ήδη πρέπει να σα πω ότι κάναμε πάρα πολύ μεγάλε και σκληρές πραγματεύση σε ό,τι αφορά τον αρχικό προπολογισμό. Γι' αυτό λοιπόν από πλευρά μα θα ήθελα να σας πω το εξή. Και εγώ και πολλοί συνάδελφοι φαντάζομαι μαζί μου θα πολεμήσουμε για μια σωστή, πλήρη, ένα πλήρη εξοπλισμό της ε, εισαγγελία με προσωπικό, επαρκές προσωπικό. Καταρχάς, ε, δεν μπορούμε να είμαστε εν μέρη, να μιλάμε για μερική απασχόληση εντεταλμένου εισαγγελεί. Και στην Eurojust είχαμε διευκρινίσει αντίστοιχα στοιχεία ότι δεν μπορεί φυσικά να υπάρχει άγνοια των εθνικών διαδικασιών, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω να μειώσουμε περαιτέρω τις δυνάμεις ε, της εισαγγελία με την ε, άσκηση καθηκόντων στις εθνικές ε, αρμοδιότητες. Γιατί αν κάποιος τελικά μπορεί να απασχολείται κατά ένα τρίτο, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πώς είναι δυνατόν να υποβάλει ερωτήματα σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τις νομοθεσίες για το ΦΠΑ της εθνικής της αρμοδιότητας και επικράτειας. Θεωρώ ότι είναι αδύνατον. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω το εξή. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να μην αποτελεί υπηρεσία, να αποτελεί ένα ευρωπαϊκό θεσμό και να έχει διαφορετικό καθεστώς. να μην ε, προέρχονται οι πορεία από το Γενικό Προπολογισμό και να εξαρτάται λοιπόν από την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή. Θα σας ευχαριστήσω επίσης που θέλετε να συμπεριλάβετε το θέμα της ε, φοροδιαφυγής σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ. Γιατί όταν κοιτάμε πραγματικά τα πόσα τα οποία χάνουμε, μιλάμε για εκατοντάδες ε, δισεκατομμύρια. Και άρα τα 3, 4, 5 δισεκατομμύρια τα οποία συζητάμε εδώ πέρα τόσο εξαρτητικά πραγματικά με αγανακτούν. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Ναι, ναι, ναι. Α, ε, ε, συγγνώμη, λέει κυρία Χολμάιρ, δισεκατομμύρια είπα, εκατομμύρια εννοούσα. Ναι, ναι, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Τα εκατομμύρια λοιπόν που συζητάμε εδώ, ενώ συζητάμε για εμ, απώλεια εσόδων σε ύψος δισεκατομμυρίων σε ό,τι αφορά το εργανομένο έγκλημα, υπάρχουν και άλλα κράτη που κάθονται και προσμετρούν τι δαπανούν σε έρευνες και τι έσοδα τελικά αποφέρει αυτή η έρευνα. Δυσκολεύομαι λοιπόν να το κοιτάξω έτσι και πραγματικά σας ευχαριστώ και θα σας υποστηρίξω. Και τώρα αν δεν κάνω λάθος κύριε Ράντεφ, τώρα προβλέπονται οι συντονιστές. Να πάρουν το λόγο οι συντονιστέ, να ξεκινήσουμε από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και μετά να συνεχίσουμε με την Επιτροπή ΚΟΝΤ. Τι προβλέπετε ακριβώς ως προς τη διαδικασία. Σε ευχαριστώ, Μόνικα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συντονιστές των δύο επιτροπών, ΛΥΜΠΕ και ΚΟΝΤ, πρώτα στους συντονιστές της ΛΥΜΠΕ και κατόπιν στους συντονιστές της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Και τους θέλω παρακαλώ να μην ξεπεράσουν το δίλεπτο στις αγορεύσεις τους, γιατί έχουμε ένα μακροσκελή κατάλογο μιλητών. Ο κύριος Λέναρς. Σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε Χαιρόμαστε ιδιαίτερος που επιτέλους φαίνεται να περνάει σε μια πιο λειτουργική φάση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ κατάγομαι από την Ολλανδία που αρχικά δεν είχε προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και χαίρομαι που ιδιαίτερα τελικά αποφασίσαμε να το κάνουμε. Αυτά που είπατε μας βρίσκουν σύμφωνος. Θέλουμε ένα μια πραγματικά ανεξάρτητη και αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όχι μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόνο όνομα. Θέλουμε πραγματικά να είναι ένα όργανο που θα αποφέρει απτά θετικά αποτελέσματα. Θέλουμε να προστατεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντα και όπου εντοπίζεται απάτες ή κακή διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων να αναλαμβάνεται δράση. Έχω δύο ερωτήσεις κυρία Κοντρούτσα. Σε ό,τι αφορά το σύστημα διαχείρισης των υποθέσεων που θα θεσπιστεί, είπατε ότι θα το ενημερώσετε. Υπάρχει επαφή Ευρωπαϊκής Αγγελίας και Eurojust, ώστε η επικαιροποίηση να γίνει προς αμοιβαία, με αμοιβαία σε τρόπο. Πώς βλέπετε τη διάρθρωση συνεργασίας Ευρωπαϊκής Αγγελίας και Eurojust στο μέλλον. Πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε μια υπόθεση με γεωργικές επιδοτήσεις, ένα μεγάλο σκάνδαλο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε στην ουσία κάτι, ότι είναι κάτι που θα πρέπει να το διερευνήσουμε περαιτέρω. Αλλά δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Φαντάζομαι στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι επιφορτισμένη με τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν κακή διαχείριση, κακή χρήση, απάτη σε γεωργικές ή άλλες επιδοτήσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τέτοιες υποθέσεις στο μέλλον, πού βλέπετε το ρόλο και τη θέση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Σας ευχαριστώ και καλή σας τύχη. Η ε, κυρία Ζήπελ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Κοντρούτσα και ο Βεσί για την παρουσίασή της και συμφωνούμε απόλυτα ότι η καταπολέμηση της απάτης και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης είναι θέμα ιδιαίτερα προσφυλές στους Ευρωπαίους πολίτες για δύο λόγους. Καταρχήν μιλούμε για κονδύλια, για χρήματα των ίδιων των φορολογουμένων. Και δεύτερον, είναι θέμα εμπιστοσύνη στι στις αρχές και στους αρμόδιους φορείς. Γιατί αν ε, δεν τηρούνται οι κανόνες από τους αρμόδιους φορείς, γιατί να τους τηρούν σε τελική ανάλυση οι πολίτες τους κανόνες. Είναι θέμα αξιοπιστής λοιπόν των θεσμών. Έχω μερικές ερωτήσεις, δεν ξέρω αν μπορείτε να τις απαντήσετε. Όταν μιλάτε για εισαγγελείς μερικής απασχόλησης, πραγματικά είναι γελίο να μιλάμε για εισαγγελείς μερική μερικής Για ποιους λόγους κάποια είναι απρόθυμα ως προς το θέμα αυτό. Γιατί διστάζουν να διεκπαιρεώσουν κάποιες έρευνες και ανακρίσεις. Μήπως σε πολλές από τις χώρες μας τα συστήματα δεν είναι αρκετά καλά εξοπλισμένα και έχουμε πραγματικά φαφούτιδες εισαγγελείς ξεδοδιασμένους χωρίς καμία εξουσία, μόνο κατόνομα. Mm. Αλλιώς ε, δεν βρίσκω λόγο, γιατί να μιλούν, έστω και να μιλούν για μερική απασχόληση αγγελή. Είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο, γιατί είναι ε, εμφανέ ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Έχω ερωτήσεις για διάφορες, για τον αριθμό των ερευνών. Σίγουρα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις απάτης ή κακής χρήσης ή κακοδιαχείρισης ε, φάνηκε και από τον αριθμό των υποθέσεων που χειρίζεται η ΟΛΑΦ. Πώς εξηγείτε εσείς ότι τώρα έχουμε πολύ περισσότερες περιπτώσεις απατώνοντας στα και κακής διαχείρισης από αυτές που αρχικά προβλέπαμε. Πώς εξηγείτε αυτή την αύξηση του αριθμού. Ευχαριστώ κύριε Ιντφέλτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την εισαγγελέα μας που ήρθε στη συνεδρίαση και την ευχαριστώ θερμά για την ε, εντιμότητά της. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτά τα αρχικά στάδια, στην αρχική φάση λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Αγγελία. να είστε σαφεί, ειλικρινεί, έντιμοι και ξεκάθαροι για τις ανάγκες του οργάνου αυτού. Και βλέπω το... Ε, τη συμπεριφορά των κρατομέλων. Το είδαμε και με το Frontex. Στην αρχή ήταν αναφανδόν ε, υπέρ του Frontex, με πλήρες αρμοδιότητες αλλά δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους στα κράτη-μέλη. Το βλέπουμε και εδώ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μπορεί να ακούγουμε κοινική, αλλά πραγματικά αρχίζω και αναρωτιέμαι αν όντως τα κράτη-μέλη θα, μήπως θα υπονομεύσουν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει από την αρχή, ότι μήπως δεν υποστηρίξουν τα κράτη-μέλη επαρκώς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και αναρωτιόμαστε και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί για να σα στηρίξει και να σα βοηθήσει. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει τι προτάσεις για τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Αγγελία και θα δώσει μάχη για τη σωστή στελέχωση και χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Αγγελία. Η κυρία Χολμάιερ είπε ότι ουσιαστικά μπαίνει η Ευρωπαϊκή Αγγελία σε άλλο τμήμα του προπολογισμού. Δεν μπορώ να κρίνω τα στοιχεία που μας δίνετε, αλλά είναι τεράστιος ο αριθμός των υποθέσεων. Μιλούμε για χιλιάδες περιπτώσεις. Οπότε, αν το πρόβλημα του δυναμικού στον ικανοτήτωτα δεν λυθεί γρήγορα, τι θα συμβεί με την ε, διαλεύκανση αυτών των υποθέσεων. Και ε, διαρωτόμαστε τι δυνατότητα επιρροή έχουμε ε, στα κράτη-μέλη για να επιταχύνουν τις ενέργειές τους. Μπορούμε να το ζητήσουμε ευγενικά μία-δύο φορές, αλλά αν εξακολουθούν να κολλησιεργούν, ίσως θα πρέπει να είμαστε κι εμείς πιο αποφασιστικοί, ε, να κάνουμε και δημοσιονομική απεργία γίνεται, να μην προχωρήσουμε στην έγκριση του προϋπολογισμού ως μέσο πίεσης ε, στα κράτη-μέλη. Οπότε, αν δεν τηρήσουν τις υποσχέσεις τους στα κράτη-μέλη και μάλιστα γρήγορα, γιατί αν δεν ξεκινήσει από την αρχή καλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα αποτύχει. Ευχαριστώ. Ποιος είναι εκπρόσωπος των Πρασίνων, συντονιστής των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών από την ομάδα μου. Ευχαριστώ κυρία Κοντρούτσα για την παρουσίασή σας και σίγουρα το νοσιακό δίκαιο δεν θα πρέπει να είναι μόνο στα χαρτιά, θα πρέπει να εφαρμόζεται και όλα, αλλιώς δεν ε, έχει νόημα. Θέλουμε απόλυτη ασφάλεια και απόλυτη υλοποίηση και συμμόρφωση και για τα φορολογικά και για το ΦΠΑ Θέλουμε αποτελεσματικές ε, ανακρίσεις και έρευνες ε, εφόσον διαπράτεται αδίκημα. Και δεν μπορούμε να δεχθούμε υποστελέχωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και υποχρηματοδότηση. Είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο. Και ευχαριστώ που το επισήμανε και η Σοφία Ιντβέλ. Θα πρέπει να βρούμε αποτελεσματικά μέσα και πίεση προς τα κράτη-μέλη για να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εφοδιάσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με το κατάλληλο προσωπικό και τον προϋπολογισμό ώστε να ανταπεξέλθει στο έργο του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για δώσω μας είπε για την κατάσταση των πραγμάτων στην υπηρεσία. Εμείς θεωρούμε ότι μπορεί σε επιχειρησιακό επίπεδο να χρειάζεται να πιέσετε αλλά ακολουθήσαμε αυτή τη μακρά διαδρομή για τη συγκρότηση της υπηρεσίας σας. Οπότε ε, τελικά όμως αυτό που κάνετε είναι να αφαιρείτε εθνική κυριαρχία από τα κράτη-μέλη και έχετε πάρα πολύ ευρείες αρμοδιότητες. Καπελώνετε τα κράτη-μέλη και παρεμβαίνετε σε αποκλειστικές αρμοδιότητες, δηλαδή στο ποινικό ε, δίκαιο. Εμεί είμαστε κατά και θα πρέπει να σας πω πω βέβαια για να μην έχουμε παρεξηγήσει ότι φυσικά και τα πρέπει να τα οικονομικά συμφέροντα και επίση να δώσουμε προτεραιότητα στην δίωξη αυτών των εγκλημάτων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Αλλά αυτό είναι αρμοδιότητα εθνική. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να διαχωριστεί από την εθνική κυριαρχία. Επομένω, μόνο εθνικέ αρχέ και με στενή δικαστική συνεργασία και με ανταλλαγή πληροφοριών ε, που είναι αρμόδιες για δίωξη της διαφθοράς. Έτσι να καταπολεμούνται αυτά τα εγκλήματα. Δεν μπορεί να έχουμε εδώ επικουρικότητα και να σας πρικοδοτεί ε, ο δημόσιος κορβανάς και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Θέλουμε να υποστηρίζουμε τις αγγελίες, θέλουμε να υπάρχει υποδομή και να δημιουργείται και επασχόληση για τους ε, νέος, γιατί ακριβώς έτσι σκέφτηκαν οι χώρες που δεν θέλησαν να συμμετάσχουν στην ε, εισαγγελία. Γι' αυτό και υπάρχουν διάφορα ε, κενά στον κοσμό λειτουργίας σας και επίσης έχουμε δει κάποια προβλήματα δομικού χαρακτήρα που αυτά προέκυψαν και Επομένως, δεν έχετε τη δομή που χρειάζεται για να λειτουργήσετε εύρυθμα. Τελικά όλα θα εξαρτηθούν κατά πόσον μπορούν να συμμετάσχουν τα κράτη-μέλη, να σας δώσουν ανθρώπινους πόρους, όπως είπατε. Όμως ε, έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν θα υπάρχει εμπιστοσύνη όσον αφορά την υπηρεσιακή σας ε, δυνατότητα. Επόμενος και ο Μποκατσίνη. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε, λέει ο κύριος Προκατσίνη. Ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα εδώ γιατί μας μιλήσατε με ευθύτητα, με ειλικρίνεια, η οποία δεν είναι συνηθισμένη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και είναι γνωστό ότι η δική μας πολιτική ομάδα ε, είχε πολλές επιφυλάξεις όσον αφορά ε, την συγκρότηση αυτού του νέου θεσμικού οργάνου της ε, Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και αυτό γιατί εμείς είμαστε προσελωμένοι σαν αρχή της επικουρικότητας επίσης. Εφόσον ο κανονισμός λειτουργίας σας τώρα είναι δεδομένος και είσαστε στη διαδικασία της ε, στελέχωσης συγκρότησης, ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο πια παρά να ευχηθούμε ότι όλα θα μπορέσουν να λειτουργήσουν εύρυθμα. Οπότε θα πρέπει βέβαια να έχετε ό,τι μέσα σας χρειάζονται για να λειτουργήσετε για να έχει νόημα η ύπαρξη της υπηρεσίας Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξή. Για δεν κάνω λάθος, το 18 ο πρόεδρος ε, Γιούγκερ θέλησε διεύρυνση των ε, αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και να καλύψετε και εγκλήματα σχετιζόμενα με τρομοκρατία. Οπότε εσείς πώς το βλέπετε με τις δυσκολίες δεδομένες που έχετε σήμερα σε σχέση με τον προπολογισμό μας θα μπορέσετε να κάνετε αυτή την επέκταση των δραστηριοτήτων, των αρμοδιοτήτων ή πρόκειται για ουτοπική ιδέα που θα πρέπει να καταληφθεί. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Good. Προχωρούμε στους συντονιστές. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ και σας κυρία Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω και σας κυρία Εισαγγελέα για την ε, σπουδαία ομιλία σας. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στις ερωτήσεις μας στην κατάσταση στα κράτη-μέλη και σε ό,τι αφορά στις ερευνές σας, την ιδιωτερότητά σας, γιατί κάθε φορά το πρόβλημα είναι το εξής. Σε πολλά κράτη βλέπουμε ποια είναι τα ζητήματα και ήμουνα σε μία αποστολή της Κόνς στη Σλοβακία, συμμετείχα. Και εκεί έγινε λόγος για την επιρροή της μαφίας στις κρατικές δομές και στις εγγελικές ε, αρχές. Η έρευνα δημοσιογραφική και η έρευνα του Γιάνν Κουτσιάκ, του δημοσιογράφου, έδειξε ότι οι μυστικές υπηρεσίες, οι εισαγγελικές αρχές, οι αστυνομικέ δυνάμεις, αλλά και ο Πρωθυπουργό ε, και οι Υπουργοί της Σλοβακίας ήταν εμπλεκόμενοι. Ήταν πραγματικά ε, απίστευτο. Πώς θα αποδείξετε εσείς όμως ότι είσαστε ουδέτεροι και πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα αυτό της μεγάλης επιρροής που ασκείται στις έρευνες και της διαπλοκής σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές ε, έρευνες. Γιατί ξέρουμε ότι το πρόβλημα με, τα ευρωπαϊκά, με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Κανείς όμως δεν ήθελε να γίνει σωστή έρευνα και δεν έγινε για πολλά χρόνια. Μέχρι ότου δολοφονήθηκε ο δημοσιογράφος και τότε ξεκίνησαν πραγματικά οι έρευνες. Αυτή λοιπόν η πολύ σημαντική ερώτηση έχω να σας απευθύνω. Θέλω να μου πείτε τι προτίθεστε να κάνετε σε ό,τι αφορά την κατάσταση αυτή και πώς θα την διαχειριστείτε με την ομάδα σας. Ευχαριστώ. κυρία Κινίτσι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Εισαγγελία που ήρθατε να μας μιλήσετε σήμερα σας ευχαριστώ που ε, τόσο ξεκάθαρα με τόση διαφάνεια μας είπατε τι ανάγκες έχει η υπηρεσία σας τόσο ώστε να αρχίσει τη λειτουργία σας. Είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα και ανθρωπίνων ε, πόρων. Νομίζω ότι πρέπει να υποστηριχθούν τα αιτήματά σας. Ε, εγώ έχω προσωπική και οικογενειακή ε, εμπειρία αλλά και από τη χώρα μου και είναι πάρα πολύ βασική η εύρυθμη λειτουργία της αγγελίας για να καταπολεμηθεί το έγκλημα και είμαι πεπισμένη ότι και εσείς θα έχετε πολύ σημαντικό ρόλο ε, για να καταπολεμήσετε και το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα που όσο περισσότερο ε, καταπολεμείται ε, αυτού του είδους η δραστηριότητα τόσο καλύτερα είναι για το ξέπλυμα, για το ξέπλυμα χρήματος, για ε, την διαφθορά που πρέπει να καταπολεμηθούν. Οπότε θα είσαστε πολύ ε, σημαντικοί σε αυτή την προσπάθεια. Οπότε, επαναλαμβάνω, χρειάζεται συγκεκριμένα να υπολογιστεί σε μέσα και ανθρώπινους πόρους τι χρειάζεστε και αυτό να καλυφθεί το αίτημα. Επίσης, σε σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες εμείς μόνο 1% έχουμε ανακτήσει από να δικαιολόγει το πλουτισμό ε, των εγκληματιών. Εσείς τι νομίζετε, ότι έχουμε νομοθετήματα σήμερα ε, τα οποία να επαρκούν ούτω ώστε να μπορέσουμε σε αυτό το επίπεδο να καταπολεμήσουμε τις ε, εγκληματικές οργανώσεις. Και αναφέρομαι στην οδηγία για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που εγκρίθηκε στην προηγούμενη θητεία. Επαρκεί αυτό ή χρειάζεται κάτι παραπάνω από πλευράς ε, νομοθεσίας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Τουγκάροφ, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και την εισαγγελία για την παρουσίαση που μας έκανε. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω. Μία για σας που έχει να κάνει με την μεγαλύτερη παροχή ε, στοιχείων. Έχετε πιο πολλά αριθμητικά στοιχεία. Τι γίνεται σε όλη την, ε, το σύστημα διαχείρισης ε, υποθέσεων. Τι σας λείπει, τι χρειάζεστε. Δώστε μας συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Υπάρχουν άλλα τμήματα όπου χρειάζεστε ενίσχυση, πού χρειάζεστε πιο πολλά χρήματα, πού χρειάζεστε πιο πολύ προσωπικό. Όσο πιο λεπτομερεί πληροφορίε γίνεται, γιατί νομίζω ότι αυτέ οι πληροφορίε θα μα επιτρέψουν να καταλάβουμε πιο καλά τι ανάγκε τη υπηρεσία. Και μία ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι στο Προεδρείο, κάπου πίσω φαντάζομαι είναι. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία για να επιληθεί αυτή η κατάσταση και για να φροντίσουμε σωστά τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν νομίζω ότι χωράνε άλλε πολιτικέ συζητήσει. Είμαστε σε μια πολύ περίπλοκη και σύνθετη κατάσταση. Δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε τα σωστά αποτελέσματα και να έχουμε μια σωστή υπηρεσία αν συνεχίσουμε να παίζουμε με τη χρηματοδότηση. Πραγματικά θα πρέπει να υπάρξει δραματική αλλαγή σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Και ρωτώ, μέχρι πότε λοιπόν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι γνωρίζουμε παρκώ και πλήρω τι χρειάζεται για τη νέα χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία. Εβδομάδε, πείτε μου, συγκεκριμένα. Πότε θα έχουμε μια μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκρίνεια σε σχέση με την κατάσταση. Πότε θα αρχίσουμε να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με σωστενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη ε, τον καθορισμό του προπολογισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και Ευχαριστώ. Η αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θεωρώ ότι μεταξύ άλλων θα αποδειχτεί από το κατά πόσο θα λειτουργήσει σωστά και εύρυθμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ξέρουμε ότι πολλές χώρες συνδέουν και πολέμησαν εξ αρχής ε, κατά της εισαγγελίας και το πρόσωπό σας ε, συγκεκριμένα ε αλλά επιμείναμε και θεωρούμε ότι είναι τεράστιο επίτευγμα αυτό που πετύχαμε. Τώρα, αυτά τα κράτη-μέλη προσπαθούν μέσω της πίσω οδού να αποδυναμώσουν, να υπονομεύσουν και να ακυρώσουν ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να αποστέλουν, για παράδειγμα, εισαγγελίε μερική απασχόληση. Απόλυτη νοησία. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό για μα ω Κοινοβούλιο να φροντίσουμε να υπάρχει σωστό εξοπλισμό με το προσωπικό που χρειάζεται η εισαγγελία. Και συμφωνώ με την Μόνικα, αυτό δεν μπορεί να είναι ει βάρο τη Όλαφ και άλλων θεσμικών οργάνων που ήδη έρχονται και παραπονιούνται. Γιατί λόγω του Brexit και λόγω της μελλοντική αύξηση του ΦΠΑ τα οικονομικά εγκλήματα τα οποία είναι προβλέψιμα και τα οποία θα του αναποστολή και απόσπαση μεγαλύτερου όγκου προσωπικού δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Η δική μα λοιπόν απέτηση θα πρέπει να είναι να υπάρξει καθαρή αύξηση του προσωπικού και του προπολογισμού. Δεν μπορεί τελικά ο καθαρό ε, προπολογισμό να είναι αρνητικό. Και αυτό θα είναι εις βάρος των ευρωπαϊκών οργάνων. Γι' αυτό λοιπόν ρωτώ, είπατε άλλωστε ότι μιλάμε για 30 έως 50 δις και το Brexit θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες παραδιάσεις και απάτες σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ. Πώς θα εκτιμούσατε λοιπόν το νέο αυτό ποσό το οποίο θα προκύψει. Κάτι άλλο το οποίο επίσης αναφέραμε, το θέμα της κατάχρησης των ε, γεωργικών ε, επιδοτήσεων και των επιδοτήσεων σε ό,τι αφορά τον τομέα των διαρθρωτικών ταμείων. Εδώ το ερώτημα που ανακύπτει είναι το εξή. Αν κάποιε χώρε δεν διαθέσουν, όπως ζητήσαμε συγκεκριμένα, πιο πολλούς εισαγγελεί, κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να συνδεθεί με τα οικονομικά του συμφέροντα από τα γεωργικά και τα διευθυντικά ταμεία. Εμεί, ως Κοινοβούλιο, το είπε και η Σοφή, τι μόχλευση μπορούμε να ασκήσουμε, πώς μπορούμε να επηρεάσουμε πιο πολύ αυτά τα κράτη-μέλη. Μήπως ε, τίθεται θέμα προπολογισμού και μήπως από εκεί θα μπορούσαμε να παρακρατήσουμε πόρους. Θεωρούμε ότι οι εισαγγελίε μερικής απασχόλησης δεν αποτελούν λύση. Δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν λύση. Χρειαζόμαστε μια σωστή στελέχωση τη εισαγγελία και είπατε ότι σε τελική ανάλυση δεν ξέρουμε καν πόσε υποθέσει θα προκύψουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα φροντίσουμε να μπορέσει να πετύχει η υπηρεσία και το κάθε κράτο μέλο. Ευχαριστώ πολύ. Για την ταυτότητα και δημοκρατία έχουμε συντονιστεί από την ΚΟΝΤ. Όχι. Οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Κέβεση για να απαντήσει στον πρώτο γύρο των ερωτήσεων των συντονιστών των δύο επιτροπών. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για τη θερμή υποστήριξή σας για το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και σας ευχαριστώ για τα ενθαρρυντικά και ψυχωτικά σας λόγια. Θα επιχειρήσω να απαντήσω εν συντομία σε όλες τις ερωτήσεις. Αν κατάλαβα καλά, η πρώτη ερώτηση αφορούσε τη συνεργασία μας με τη Eurojust. Σας διαβεβαιώ ότι ήδη έχω επαφές με τον πρόεδρο της Eurojust. Ήδη έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές και αρχίζουμε, αρχίσαμε τη διαπραγμάτευση των, της εργασί, των εργασιών και της συνεργασίας μας. Πρώτα σε, σε τεχνικό επίπεδο, αλλά όλες ε, οι ρυθμίσεις ε, συνεργασίας θα πρέπει να ε, εγκριθεί από το κολέγιο των εισαγγελέων. Προς το παρόν δεν έχει σταθεί, οπότε έχει παγώσει η διαδικασία. Από τη στιγμή που θα διοριστούν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, θα συσταθεί το συλλογικό όργανο και θα δούμε τι συνεργασία τεχνική θα έχουμε με τη Eurojust. Και προσελεύουμε σε στενή συνεργασία με τη Eurojust, γιατί είναι σημαντική τεράστια εμπειρία που έχει το όργανο αυτό με τη διεθνή συνεργασία, αλλά θα πρέπει να έχουμε στενή συνεργασία και με την Europol και την Olaf και όλες τους άλλους ε, ευρωπαϊκούς οργανισμούς ή φορείς. Τώρα, ε, δεν μπορώ να σας αναλύσω τις λεπτομέρειες, γιατί δεν θα τις καθορίσω εγώ τις λεπτομέρειες συνεργασίας με την Eurojust, αλλά το συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τώρα, πώς θα ε, διερευνηθεί η χρήση των γεωργικών κονδυλίων. Θα κάνουμε ίδια, ίδιο τρόπο έρευνα ε, με οποιαδήποτε άλλη κακή διαχείριση, κακή χρήση κονδύλιων. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχουμε ακόμη αρχίσει τι δραστηριότητε, δεν μπορούμε να μιλάμε για έρευνε. Σε ό,τι αφορά το θέμα των ε, εισαγγελέων μερική απασχόληση, θα σα διαβεβαιώ ότι καθ' όλη τη σταδιοδρομία μου δεν είδα μισό εισαγγελή ή ένα τέταρτο εισαγγελέα. Μερική απασχόληση εισαγγελή δεν έχω ακούσει ποτέ. Και αν δεν έχουμε πλήρου απασχόληση στις αγγελίες, δεν μπορούμε να, εγγυηθούμε ούτε την ανεξαρτησία τους, ούτε την ευθύνη τους, ούτε την αποτελεσματικότητά τους. Θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρε αρμοδιότητες και να είμαστε αποτελεσματικοί. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τις πλήρου πλήρους απασχόλησης. Και ελπίζω ότι στι διαπραγματεύσει που έχουμε ξεκινήσει με όλα τα κρατη ε, θα καταφέρουμε να επιτύχουμε τη συμφωνία τους για εισαγγελείς πλήρους απασχόλησης. Είναι πολύ σημαντικό να ευοδοθούν οι συνομιλίες με τα κράτη-μέλη στο θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα την αξιολόγηση της νομολογίας, σε μια προκαταρκτική αξιολόγηση που έκανα, έλαβα υπόψη αντικειμενικά κριτήρια και κυρίως τις απαντήσεις που έλαβα από τα κράτη-μέλη για τις υποθέσεις που διερεύνησα τα κράτη-μέλη την τελευταία τετραετία και ζήτησα τα στατιστικά στοιχεία μόνο για τις υποθέσεις που βρίσκονται υπό την δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής αγγελίας. Με βάση τις απαντήσεις που έλαβα από τα κράτη-μέλη έκανα κάποιες προκατακτικές αξιολογήσεις και υπολόγισα ότι από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας θα λάβουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περίπου 3.000 υποθέσεις. Και με βάση τις πληροφορίες αυτές διαπιστώνω ότι κάθε χρόνο οι νέες υποθέσεις που φτάνουν στα εισαγγελικά γραφεία είναι περίπου 2.000. 2.000 το χώρο, το χρόνο. Οπότε ήδη την πρώτη μέρα θα λάβουμε 2.000 υποθέσεις και κάθε χρόνο θα, λαμβάνουμε θα αναλαμβάνουμε και 2.000 νέες υποθέσεις. Αυτό υπολόγισα. Δεν ολοκλήρωσα όμως την αξιολόγηση του αριθμού των υποθέσεων, γιατί δεν έχουν στείλει ακόμη όλες οι χώρες μέλη τα στατιστικά στοιχεία. Οπότε δεν μπορώ να είμαι κατηγορηματική στα συμπεράσματά μου. Θα λάβω τα στοιχεία και θα ε, αξιολογήσω κατά πόσο εμπίπτουν στην δικαιοδοσία μας υποθέσει υποθέσεις αυτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημα τι θα συμβεί ε, με την διεκπαιρέωση των Υποθέσω σε περίπτωση που δεν έχουμε επαρκή στελέχωση ή επαρκή προπολογισμό. Μα δεν μπορούμε να αναλάβουμε δραστηριότητε αν δεν έχουμε επαρκέ προσωπικό και προπολογισμό, γιατί υπάρχει κίνδυνο να κολλήσουν οι δραστηριότητέ μα. Και θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Α υποθέσουμε ότι φέτο θα ξεκινήσουμε τι δραστηριότητε με 29 μέλη προσωπικού, 22 εντεταλμένου εισαγγελεί και 32 29 συγγνώμη εισαγγελείς και 32 ε, εντεταλμένους εισαγγελείς. Ήδη στο Λουξεμβούργο 25 ε, υπάλληλοι έχουν αποσπαστεί για ανθρώπινους πόρους, για IT, τεχνολογία των πληροφοριών και για δημοσιονομικά θέματα. Θέλουμε προσωπικό και σε αυτούς τους τομείς. Αλλά για το επιχειρησιακό σκέλος έχουν απομείνει μόνο τέσσερις υπάλληλοι. Είναι πολύ δύσκολο με τέσσερις υπαλλήλους να κάνουμε καταγραφή και ανάλυση 3.000 υποθέσεων που υπολογίζουμε ότι θα λάβουμε μόνο με τέσσερις υπαλλήλους που έχουν απομείνει για τα επιχειρησιακά θέματα, για το επιχειρησιακό σκέλος, αφού οι άλλοι είναι αποσπασμένοι ε, στα δημοσιονομικά και άλλα θέματα. Επίσης, Κάποιο ρώτησε αν γίνεται επέκταση ή παράταση της εντολής για να καλύπτει και εγκλήματα τρομοκρατία. Νομίζω ότι είναι πρόωρη η συζήτηση για τα θέματα αυτά. Είπα ήδη το Δεκέμβριο στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών να δούμε αν θα ξεκινήσει σωστά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πώς θα λειτουργεί και εν πάση περιπτώσει δεν είναι δική μου απόφαση αν θα παραταθεί η εντολή του ΕΠΟ, αν θα γίνει η διεύρυνση τη εντολή για να καλύπτει και άλλα εγκλήματα στη δικαιοδοσία του. Η νομοθετική εξουσία θα αποφασίσει, οι νομοθέτε. Σε ό,τι αφορά τι ερωτήσει τη Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, για το πώ θα, εξασφαλίσουμε και θα εγγυηθούμε την ουδετερότητά μα σε ό,τι αφορά την έρευνα στα κράτη-μέλη. Η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η ανεξαρτησία των εισαγγελέων του γραφείου μας εξασφαλίζεται τον ίδιο τον κανονισμό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι ανεξάρτητη. Αυτό είναι ένα στοιχείο απαραίτητο που κατοχυρώνεται στον κανονισμό. Και, και στην οργάνωση του Ευρωπαϊκού Εισαγγελε... του, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουμε, έχουμε και μόνιμα τμήματα που παντρώνονται από τρεις εισαγγελίες από διαφορετικά κράτη-μέλη. Και μόνο για αυτή την οργάνωση μπορούμε να πούμε μια ανεξαρτησία κάθε υπόθεσης και κάθε έρευνα θα εξασφαλίζεται. Γιατί όλες οι έρευνες που θα γίνονται από τους εντεταλμένους εισαγγελείς στα κράτη-μέλη τους αλλά θα εποπτεύονται από τα μόνιμα τμήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και θα έχουμε τρεις διαφορετικούς εισαγγελείς από τρία διαφορετικά κράτη-μέλη σε αυτό το μόνιμο τμήμα. Επίσης, μπορούμε να εγγυηθούμε την ανεξαρτησία και την ουδετερότητα των ε, ερευνών, καθορίζοντας ε, κάποια αντικειμενικά κριτήρια για το, την ανάθεση των υποθέσεων και την ανακατανομή ενδεχομένω των υποθέσεων. Αυτό θα το αποφασίσει το Συλλογικό Όργανο της Ευρωπαϊκής, Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Τώρα, για το πώς θα καταπολεμήσουμε ε, κάποια τέτοια εγκλήματα και με τι μέσα. Δεν ξέρω αν έχουμε όλα πια τα εργαλεία για να τα αξιοποιήσουμε όλα. Είναι πολύ νωρίς να πούμε αν, χρειαστούμε, αν θα χρειαστούμε και νέο εργαλείο ή νέο μηχανισμό. Ούτε είναι δική μου αρμοδιότητα να πω αν κάποιες οδηγίες ή κάποια νομοθετικά μέσα θα πρέπει να τροποποιηθούν. Επίσης, στέθηκε μία ερώτηση για το πού χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους και κονδύλια. Όπως είπα, ολοκλήρωσα μία προκαταρκτική αξιολόγηση, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο, γιατί ακόμη δεν έχει σταθεί το συλλογικό όργανο των εισαγγελέων και λόγω του δημοσιονομικού χρονοδιαγράμματος ε, οφείλαμε να στείλουμε μία πρόταση. Οπότε έκανα αυτή την προκαταρκτική αξιολόγηση και την υπέβαλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έστειλε επιστολές στους επιτρόπους και το μπαλάκι τώρα είναι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκείνη θα υποβάλει την πρόταση του προπολογισμού για το ΕΠΟ. Και μετά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι συνομοθέτε θα αποφασίσουν για το ύψο αυτού του προπολογισμού. Σε ό,τι αφορά τι απώλειε από τις απάτες ΦΠΑ. Έχουμε τη μελέτη ΚΕΛ και κάναμε Ε, την ανάλυση των εισαγωγών-εξαγωγών στο διμερές εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι διαφορές ε, στις, ε, στα στοιχεία εξηγούνται από τις απάτες ΦΠΑ και οι υπολογισμοί της μελέτης αυτής για, τις, για την απάτη είναι μεταξύ 30 και 50 δις. Και δεν ξέρω πώς το Brexit θα επηρεάσει το ύψος αυτής της ζημίας από την μη καταβόλη ΦΠΑ, η μελέτη δεν κατονομάζει συνήθεις υπόπτους, θεωρεί ότι είναι ζήτημα κοινό σε όλα τα κράτη-μέλη η απάντηση στο ΦΠΑ. Νομίζω ότι απάντησα. Και αν έχετε και άλλες απορίες, παρακαλώ να τις ακούσω. Περνάμε τώρα στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Είναι μεγάλος ο κατάλογος. Να ζητήσω λοιπόν από τους συναδέλφους να περιοριστούν στο ένα λεπτό, εφόσον είναι δυνατόν. Και μετά να ακούσουμε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Γιάννη εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να σας ευχαριστήσω και για την αποφασιστικότητά σας. Να πατύχετε αποτελέσματα ανεξαρτήτως του προπολογισμού σας, όπως είπατε δουλειά και η εργασία της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας θα εξαρτηθεί και από τη συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Πώς θα εξασφαλίσετε λοιπόν την πραγματική ανεξαρτησία της ε, των Ευρωπαίων ε, ενταλμένων εισαγγελέων και πώς θα διεξαγάγετε ανεξάρτητες ερευνές με υψηλό σε ό,τι αφορά υψηλό βαθμού αξιωματούχου. Σε ό,τι αφορά την Europol. Πώ φαντάζεστε ότι θα σα υποστηρίξει στι μελλοντικέ σα εργασίε και στι ερευνέ σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Κουλακούσιτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Κοβέζη. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Πέρα από την απάτη σε σχέση με το ΦΠΑ, πολλές ε, ε, μελέτες ε, καταδεικνύουν ότι χάνουμε στο επίπεδο αυτό δεκάδες ε, ε, εκατομμύρια στην απάτη, στην διαφθορά. Χάνουμε λοιπόν... Που βλάπτουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Εμείς τώρα έχουμε μοναδική ευκαιρία. Έχουμε το καλύτερο δυνατό πρόσωπο ε, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής ε, εισαγγελία. Η κυρία Κοντρούτσα απέδειξε πόσο ικανή είναι να πατάσει τη διαφθορά και στην πατρίδα της. Δεν θα πρέπει να χάσουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε κατάλληλο προϋπολογισμό. Και με λίγα μέσα θα μπορούσαμε να ανακτήσουμε δισεκατομμύρια στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και να επιστρέψουμε και στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε συνεπείς και να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα μέσα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ, κυρία Εισαγγελέα. Θα ήθελα, όπως και οι συνάδελφοί μου, να σας ευχηθώ ότι καλύτερα και να σας εκφράσω την υποστήριξή μας για την αποστολή σας, την οποία την αναμένουν όλοι οι Ευρωπαίοι που θεωρούν ότι η καταπολέμηση της απάτης σε όλες τις μορφές και όλες τις μορφές διαφθοράς αποτελούν ζήτημα κορυφαίο. Και πραγματικά εκφράσω το σεβασμό μου και την ε, το θαυμασμό μου για την επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Θα ήθελα να σας πω ότι η κυρία Χολμάιερ, η οποία είναι επικεφαλής του προπολογισμού με όλη την προθυμία η οποία έχει καταδείξει να σας δώσει πιο πολλούς πόρους, πρότεινε εκατομμύρια, τα οποία μπορούμε να τα ανακτήσουμε σε ό,τι αφορά τον κλάδο αυτό της δικαιοσύνης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την υποστήριξή σας και θα ήθελα να σας πω ότι σας υποστηρίζουμε αγαπητή κυρία Χολμαϊρ. Δύο ερωτήσει να σας θέσω σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Έχετε συγκεκριμένες προσδοκίες, επιθυμίες σε ό,τι αφορά την ε, διαμόρφωση της υπηρεσίας σας και κατά δεύτερον σε ό,τι αφορά το θέμα της διακυβέρνηση και της διαχείριση στη φάση της ε, κατάρτισης του μηχανισμού αυτή υπάρχει εδώ ανοιχτό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη προκειμένου να μπορέσετε να βρείτε τη θέση σα, ασφαλώ διατηρώντα και την εξαρτησία σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, και Πρόεδρο. κυρία σας ευχαριστώ πάρα πολύ. κυρία Εισαγγελέα που είσαστε εδώ σήμερα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σκληρή δουλειά που έχετε ήδη κάνει και στην προηγούμενη θέση σα από τότε που επίσημα συστάθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η καταπολέμηση τη διαφθορά και τη απάτη θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Και εμεί εδώ στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σα δώσουμε τα απαραίτητα μέσα, του απαραίτητου πόρου για να κάνετε σωστά τη δουλειά σα. Δύο ερωτήσει να σα κάνω. Καταρχά. πιστεύετε ότι θα ήταν δυνατόν τα αριθμητικά στοιχεία αυτά που μας τα προηγουμένω να δημοσιευθούν, να αναφερθεί δηλαδή Ποιε χώρε διστάζουν να βοηθήσουν το γραφείο του εισαγγελέα. ποιε χώρε είναι υπερβολικά επιβαρημένε, Θεωρώ ότι θα ήταν σημαντικό το κοινό να τα γνωρίζει αυτά. Κατά δεύτερον, φαντάζεστε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα παίξει ένα ρόλο στο μηχανισμό κράτους ε, δικαίου, αρισιμότητας κράτους δικαίου που τον κοιτάμε στον επόμενο προϋπολογισμό και επίσης θα μπορούσατε να φανταστείτε να επεκταθεί η λίστα των χωρών που υπάρχονται στην Ευρωπαϊκή Συγγελία. Έχουμε υπογραφές στην Ουγγαρία για να συμμετέχει η Ουγγαρία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη υποστήριξη από πλευρά τη χώρα μου πέρα από τα όσα αποφασίζει η κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριο Σινιέτσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την κυρία Εισαγγελέα που είναι εδώ σήμερα. Και εγώ θαυμάζω όπως οι συνάδελφοί μου το έργο σας, την αποφασιστικότητά σας και όλα όσα κάνετε για να καταστεί λειτουργική η ευρωπαϊκή συγγελία με ανεξάρτητο ασφαλώς τρόπο. Μία ερώτηση η οποία συνάδει με αυτά που είπε η κυρία Τσε. Συνεργασία σε ό,τι αφορά τις χώρες που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Συγγελία. Πείτε μας πώς συνεργάζεστε με τις κυβερνήσεις αυτές, γιατί παραδόξως, ίσως και όχι, Ξέρουμε ότι οι χώρε ε, οι οποίε δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αυτέ που αντιμετωπίζουν τα πιο πολλά προβλήματα με το κράτο δικαίου και που αντιμετωπίζουν και προβλήματα με του ευρωπαϊκού πόρου. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό. Εμένα μου φαίνεται απλά εύγολο όταν μιλάμε για ρεσιμότητα σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Μία από τι ε, συνθήκε, ένα από του όρου θα πρέπει να είναι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριο Τσουντάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ορίσατε και εσύ και από την πλευρά μα, ε, κυρία Εισαγγελέα. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την απάτη και την διαφθορά και χρειαζόμαστε λοιπόν μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κυρία Κούβεση, καταβάλλατε προσπάθειες για να ενισχύσετε τις ε, εθνικές αρχές καταπολέμησης της απάτης. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν το εξής θα καταπολεμήσετε και το, την παράνομη διακίνηση ανθρώπων διαστοριακά. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Ίσως ε, θα πρέπει να ενισχύσουμε τους Ευρωπαίους εισαγγελείς ε, για να μπορούν να ασκούν πιο αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους και τι μηχανισμό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε τα χαμένα αυτά έσοδα. Μιλάμε για μεγάλα ποσά και θα ήταν σημαντικό να ευεδεθούν τα ποσά αυτά στην ε, υγεία, στην παιδεία και σε άλλους τομείς. Ευχαριστώ πολύ και σας υποστηρίζουμε λοιπόν. Thank you. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ο επόμενος. Σας ευχαριστώ πολύ, mm. κυρία Σεγγελέα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενέργεια που έχετε δαπανίσει για όλη αυτή την ορμή που μα επιδεικνύεται γιατί μα δίνει πολύ μεγάλε ελπίδε σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη διαφθορά. Τα ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα θεωρούμε ότι θα τα προασπιστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αν η ευρωπαϊκή αυτή πόρτα, ευρωπαϊκά κονδύλια συνδεθούν με το κράτος δικαίου. Και αυτό θα πρέπει να το φροντίσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως είπε και η κυρία Τσε, η διαφθορά στην Ουγγαρία αποτελεί ένα θεσμοθετημένο κεντρικό φαινόμενο, θα λέγαμε. Οι πιο πλούσιοι Ούγγροι είναι φίλοι του Προέδρου, του Πρωθυπουργού και η οικογένειά του. Στην Ουγγαρία, λοιπόν, αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα. Ρωτώ λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να δράσουμε στις χώρες εκείνες όπου η διαφθορά είναι σε κεντρικό επίπεδο, όπου η χώρα δεν δείχνει καν οποιοδήποτε ενδιαφέρον να προσαρτηθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά προσπαθεί να την μπλοκάρει αντιθέτω. Τι μπορεί να γίνει εκεί. now for European Commission, Mr. from... Ο αρμόδιος συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Θα επαναλάβω αυτά που είπε ο ε, Επίτροπος Ρεντέρς πριν από λίγες εβδομάδες στα πλαίσια του δομένου διαλέγου είπαμε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε την Γενική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Χολμάιερ Μα συγγνώμη, δεν μου αρκούν αυτά που μα είπατε. Είναι σχεδόν προκλητική η απάντησή σα. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένω κάτι παραπάνω από μια απλή δήλωση ότι θα προβεί σε κάποιε έρευνε και ελέγχου. Δεν είναι δυνατόν να το δεχτούμε αυτό ως απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένω μία δήλωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν πρόκειται να αποδεχτεί ε, εισαγγελίε μερική απασχόληση. Θα ήθελα να ξέρω πόσες ε, θέσεις χρειάζονται ε, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πώς τοποθετείται σε όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η απάντηση πραγματικά είναι ανεπαρκέστατη. Thank ευχαριστώ. Ε, ξέρετε, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτό το θέμα και για αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει τότε να μας διαβιβάσει μια απάντηση εγγράφως, το συντομότερο δυνατόν, αφού δεν μπορείτε τώρα να απαντήσετε στα όσα θέλουμε. Έχετε τον λόγο, κυρία Συγγελέφ. Σας ευχαριστώ για τα όσα ρωτήσατε. Όπως ε, προείπα, η ανεξαρτησία της υπηρεσίας μας των εισαγγελέων, των αποσπασμένων εισαγγελέων σε σχέση με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, διεθνή ή εθνικά, ε, είναι κατοχυρωμένα από τον κανονισμό λειτουργίας. Και θα υπάρχει ένα τμήμα διαρκούς λειτουργίας όπου θα έχουμε τρεις διαφορετικούς από διαφορετικές χώρες συναδέλφους και με τους ε, υπόλοιπους συναδέλφους πρόκειται να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις με αντικειμενικά κριτήρια σε σχέση με το αν θα διεκπαιρεθούν κάποιες υποθέσεις ή αν θα διαβιβαστούν αρμοδίως. Επίσης, ε, είχαμε τις πρώτες επαφές με το Εθνές Δικαστήριο και θα πάω και με τη Europol και γι' αυτό και θα πάω σε Eurojust και Europol στη Χάγη. Οπότε και θα μπορέσουμε να αρχίσουμε τις επαφές για τεχνικά θέματα. τελικά θα ληφθούν αποφάσεις για το βαθμό συνεργασίας. Εγώ θα ήθελα να έχω στενή υπηρεσία με τις υπηρεσίες που μπορεί να Αλλά ίσως ε, αποφασιστεί κάτι διαφορετικό. Τον Ιανουάριο ξεκίνησε η διαβούλευση με τα κράτη-μέλη όσα συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 22 κράτη-μέλη. Ε, δεν έχω προλάβει ακόμη να τα επισκεφθώ όλα αυτά τα κράτη. Προσπάθησα κάθε εβδομάδα να καλύψω δύο-τρία ε, κράτη-μέλη. Και μετά τις διαβουλεύσεις θέλω να πετύχουμε τα εξής. Πρώτα-πρώτα να δούμε πώς η οδηγία, τη λειτουργία μας θα εφαρμοστεί. Δεύτερον, τι μέτρα κάθε κράτος μέλος έλαβε για να προσαρμόσει ε, στο δίκαιό του και να προετοιμαστεί για τη συνεργασία με την υπηρεσία μας και αφού μετέφερε στο ιστορικό δίκαιο τον αγωνισμό. Επίσης να δούμε τι θα γίνει με τους αποσπασμένους αγγελίες γιατί σύμφωνα με τον κανονισμό θα πρέπει αυτό να το καθορίσουμε ε, μετά την διαβούλευση το πόσοι θα αποσπαστούν από κάθε κράτος μέλος και ελπίζω ότι όλα τα κρατημέλη θα συμφωνήσουν ότι για να υπάρξουν ε, ανεξαρτησίας, ε, ευθύνης, ε, αποτελεσματικότητάς μας χρειάζονται εισαγγελείς πλήρους απασχόλησης που είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τα ίδια στάνταρ σε όλα τα κράτη-μέλη. Να μην υπάρχει πολυφωνία σε σχέση με το πώς πρέπει να λειτουργούμε. Και εννοώ τώρα και το Τη σχέση εργασία και πόσοι θα είναι οι αποσπασμένες αγγέλες. Προκρατική μου αξιολόγηση είναι αυτή για το προσωπικό και για την υπηρεκοδότηση ακόμα δεν έχει ε, συνέλθει το Συμβούλιο και έχουμε επίσης και την ομάδα εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε από μέλη όλων των κρατών που συμμετέχουν. Κάποια κρατημέλη έχουν επιφυλάξει για την υπηρεσία μας. Πάντως τώρα δεν μπορώ δημοσία να σας πω πόσες είναι οι υποθέσεις ανακράτος μέλος και πόσοι είναι οι αποσπασμένοι αγγελίες ανακράτος μέλος και πόσοι θέλουν πλήρη απασχόληση των εισαγγελίων, γιατί ακόμα είναι εν εξελίξει οι συζητήσεις, οι επαφές, οι διαβουλεύσεις. Άρα το πιο σωστό είναι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τα κράτη-μέλη, να έχουμε μία σαφή εικόνα του τοπίου, οπότε τότε να δούμε τι θα γίνει. Αλλά δεν μπορώ να σας πω τίποτα σε σχέση με τα προβλήματα ε, για κάθε κράτος μέλος για το προσωπικό, αλλά έχω ήδη κάποια στατιστικά στοιχεία, αλλά θέλω να καταλάβω γιατί έχουμε αυτά τα προβλήματα, αυτές τις ε, διαφορές από κράτος σε κράτος, μόνο όταν αρχίσουμε την λειτουργία μας. Τώρα για τον ρόλο της υπηρεσίας στον νέο μηχανισμό για το κράτος δικαίου. Νομίζω ότι η ρύθμιση που ορίζεται στον οργανισμό είναι ξεκάθαρη, οπότε τώρα θα ασχοληθούμε με έρευνες και ποινικέ διώξεις όπου ε, προβλέπεται. Δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτε άλλο. Τώρα όσον αφορά με τα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν και τι σχέσεις θα έχουμε, άρχισα όπως είπα τις ε, διαβουλεύσεις με αυτούς που συμμετέχουν στην υπηρεσία. Όταν τελειώσουν αυτή η διαβούλευση θα αρχίσω κάποιον διάλογο επικοδομητικό με τα ε, κράτη που δεν συμμετέχουν. Είναι σημαντικό να έχουμε καλή επαφή και έτσι να βρούμε ε, έναν τρόπο συνεργασίας. για αυτές τις χώρες και για άλλες. Τώρα, όσον αφορά τις έρευνες για τις χώρες που δεν συμμετέχουν, θα κάνουμε ό,τι προβλέπεται από τον νόμο σήμερα. για τον ε, Ρουμάνο βουλευτή να απαντήσω στα ρουμανικά. Όσον αφορά το δουλεμπόριο, την λαθροδιακίνηση προσώπων και την παρέκταση της αρμοδιότητας της εισαγγελίας για αυτό το έγκλημα, σας είπα ήδη είναι νωρίς να μιλήσουμε για το αν αυτό μπορεί να ρυθμιστεί. Πρόκειται για απόφαση του συνομοθέτη. Το ίδιο ισχύει και για το πόσες οι θα είναι από κάθε κράτος μέλος. Θα καθοριστεί ο αριθμός των αποσπασμένων εισαγγελέων αφού ολοκληρωθούν οι επαφές με τα κράτη-μέλη. Προσπαθούμε να έχουμε αντικειμενικά κριτήρια και όχι μόνο τις στατιστικές σε σχέση με τις υποθέσεις ανά κράτος λάβουμε υπόψη το σύστημα δικαίου κάθε χώρας και τέτοια κριτήρια. Θέλουμε να είμαστε κέντρο αριστείας. Να ξεπεράσουμε κάποιες προκαταλήψεις. Να υπάρχει ενιαία ρύθμιση. Και να Είμαστε ένας κόμβος επικοινωνίας με τις εθνικές εγγελίες. Και επίσης όσον αφορά την ανάκτηση των ε, οικονομικών ζημιών και αυτό έτσι να το ρυθμίσουμε. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε κυρία Κεβεσή. Πραγματικά ήταν πολύ διεξοδικές οι απαντήσεις σας. Η κυρία Τσέχσιτσε το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. I just wanted to comment on the previous remarks by the Commission νομίζω την επόμενη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνει εκπρόσωπο να είναι αρμόδιο άτομο για το θέμα που συζητούμε, όχι απλώς να έρχεται για να έρχεται. Αυτό ήταν ένα σχόλιο για την εκπροσώπηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να σα ευχαριστήσω καταρχά από πλευρά μα, γιατί ε, καταλαβαίνουμε από αυτά που μα λέτε πόσο σκληρά δουλεύετε και πώ καταβάλλετε προσπάθειες μαζί με όλη την ομάδα σας για να ε, στήσετε στα πόδια του την οργανισμό, την ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πόσο δύσκολο είναι το έργο σας για να σας υποστηρίξω. Ε, έχω ένα ολόκληρο κατάλογο ερωτήσεων, τον οποίο δεν καλείστε φυσικά να απαντήσετε τώρα εδώ, για να καταλάβουμε πιο καλά πού χρειάζεστε υποστήριξη. Όχι για έλεγχο, αλλά για να ξέρουμε ακριβώς πού βρίσκονται τα προβλήματα και πού βρίσκονται οι ελλείψεις, πού χρειάζεστε περαιτέρω υποστήριξη, για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και στους συναδέλφους ε, και από τις δύο επιτροπές πώς μπορούμε πραγματικά να σας ε, παρέχουμε υποστήριξη, ενίσχυση από τις ε, δύο συναρμόδιες επιτροπές και από την Επιτροπή για τον Προπολογισμό. Σας εύχομαι λοιπόν ότι καλύτερο στις μελλοντικές σας εργασίες. Σας σεβόμαστε ιδιαιτέρως και ελπίζω να πετύχετε τους στόχους σας. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας υποστηρίξουμε και στην διαδικασία αυτή των λόγο ζητάει συνάδελφος. Ε, να σας ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες και με τον κύριο Χάνο, γιατί θεωρώ ότι αυτός είναι το άτομο κλειδί, το οποίο θα μπορούσε να δώσει το πράσινο φως για να ενισχυθεί ο προπολογισμό. Ωστόσο, δεν έχει απαντήσει, δεν έχει ανταποκριθεί, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου πλέον. Μέχρι ότου δεσμευτεί πραγματικά σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη σχετική πρικοδότηση. Η κυρία Χολμάιερ. Ο Επίτροπο Χάν, από την αλήθεια, δεν είχε κάνει την ευκαιρία για να απαντήσει. Γιατί η κυρία Κούβεση μόλις τώρα υπέβαλε την έκθεση για τον αριθμό των θέσεων που χρειάζεται. Και ελπίζω να εκπληρωθούν οι, υποχρε... του Επιτρόπου Οιτιγκέρ και να μπορέσουμε να πείσουμε και τον Επίτροπο αλλά και όλο τον σώμα των Επιτρόπων ότι χρειάζεται αυτή η ενίσχυση. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Θα σας δώσω λοιπόν τις ερωτήσεις αυτές να τις πάρετε μαζί σας. Δεν ε, περιμένω άμεσα απάντηση, αλλά αν χρειάζεστε οτιδήποτε να μας ενημερώσετε και ξέρουμε, θέλουμε να ξέρουμε πόσο συνεργάζονται μαζί σας τα κράτη-μέλη, τι προθυμία καταδεικνύουν και από Επιτροπή σε Ελέγχου Προπολογισμού. Ξέρουμε ότι σε διάφορες περιστάσεις όπου όλα είχε ζητήσει τη δεξαγωγή έρευνας, ε, οι εισαγγελίε δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα αιτήματα αυτά. Τώρα λοιπόν θέλουμε να ακούσουμε, να δούμε τι θα γίνει όταν υπάρχει σύσταση για διεξαγωγή ε, ε, ελέγχων και ερευνών. Πώ θα μπορεί να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ελπίζω να συνεργαστούν μαζί σα επικοδομητικά και άκοπα όλα τα κράτη-μέλη και προκειμένου αυτή η συνεργασία τελικά να καταλήξει στην καταπολέμηση τη διασυνοριακή απάτη που υποσκάπτει τα οικονομικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ε, εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία και σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σα. Η κυρία Σίπελ. Η κυρία... Σα ευχαριστώ. Η κυρία Ιντβελτ, μάλλον. Ε, με κνεύρισε κάπως η συζήτηση σήμερα, γιατί ακούμε συνεχώς τα ίδια. Ίσως θα πρέπει το Προεδρείο και οι συντονιστές των δύο επιτροπών να συνεδριάσουν και να δουν τι μέσα έχουμε. Γιατί μπορούμε να, να ρωτάμε ευγενικά το Συμβούλιο και την Επιτροπή, αλλά μάλλον δεν θα λάβουμε απάντηση. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να συνεννοηθούν οι συντονιστές και των δύο επιτροπών να δούμε τι πίεση μπορούμε να ασκήσουμε στα κράτη-μέλη και την Επιτροπή για να ανασκουμποθούν και να αναλάβουν δράση. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντβέλτ. Νομίζω ότι ήταν πολύ καρποφόρα και εκτενή η σημερινή συζήτηση. Ευχαριστούμε κυρία Κοντρούτσα Κιόβεση. Βλέπετε ότι μπορείτε να υπολογίζετε στη βοήθεια και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο μέλλον. Και στο μέλλον ό,τι προβλήματα ανακύψουν στο έργο σα, μπορείτε πάντα να αποτείνεστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί θα το βρείτε σύμμαχο στο έργο σα. Σα ευχαριστώ και ευχαριστούμε θερμά για τη διεξοδική ανάλυση που μα κάνατε. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για το σημείο 5. Bien, nos falta un punto para terminar la sesión de hoy. έχει μείνει ένα σημείο για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή ημερήσια διάταξη. Το σημείο 6. Καθίστε παρακαλώ συνάδελφοι για να αποτελειώσουμε την ημερήσια διάταξή μας. El siguiente Επόμενο σημείο της ημερήσης διάταξης και τελευταίο αφορά ενημέρωση της Επιτροπής για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις που γίνονται επί της νομοθετικής πρότασης που θεσπίζει το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας στα πλαίσια του επόμενου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Η αρμόδια για την ενημέρωση αυτή στην Επιτροπή Λίμπη είναι η κυρία Μόνικα Χολμάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητή Μαϊτέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Με πάσα ειλικρίνεια πρέπει να πω ότι δεν βλέπω τους σκιώδεις εσύτες εδώ πέρα και δεν έχω πολλά να σας πω. Να σας ε, πω, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι να σας πω γιατί δεν έχει μειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος και αυτό γιατί να εκφράσω καταρχάς την απορία μου για το γεγονός ότι στο Συμβούλιο ε, κυκλοφορήσε η φήμη ότι δεν θέλουμε εμείς τα ως βουλευτές να διαπραγματευτούμε και να προχωρήσουμε. Αυτό που διαπιστώνω όμως είναι ότι το Συμβούλιο και οι Προεδρίες, ούτε με τη Φιλανδική Προεδρία δηλαδή, ούτε με την Κροατική Προεδρία δεν έλαβε διαπραγματευτική εντολή. Και άρα καθόμαστε ωραία ωραία. Το προσπαθήσαμε να κάνουμε και έναν τριμερή διάλογο, αλλά το πολύ πολύ να αναφέρουμε τα εντελώς αυτονόητα. Μία απλή ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών. Τα βασικά. Αλλά όλα τα θέματα τα οποία επιδέχονται διαπραγμάτευση, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει κάτι ενδιαφέρον εκεί να επισημάνουμε. Χωρίς ε, διαπραγματευτική εντολή γίνεται η σύνοδος και όπου ενδεχομένως ε, ε, να μπορούσε να συμφωνήσει το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο, εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ως νομοθέτης διαφωνεί. Φυσικά είναι, έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει ερωτήσει, αλλά δεν μπορεί να διαμορφώσει όλες τις διαπραγματεύσεις βάσει των επιθυμιών της. Ως Κοινοβούλιο φυσικά πρέπει να ακολουθήσουμε τις δικές μας γραμμές, όχι τις επιθυμίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη διατύπωση για την κουλτούρα αυτή μυστικών υπηρεσιών. Για κάποια κρατημέλη φυσικά αυτό είναι δύσκολο σε διατύπωση. Και ζήτησα από το Συμβούλιο να μας πούν πώς μπορούν να εξασφαλίσουν ότι η μελλοντική συνεργασία στο θέμα της οργανωμένης, του οργανωμένου κλίματος, στο θέμα της τρομοκρατίας, πώς θέλανε να διατυπωθεί αυτή η έννοια, αυτό το θέμα της στενής διαπλοκής, έστω να μην υπάρχει αυτή η κουλτούρα μυστικών υπηρεσιών. Αλλά δεν έχουμε ακούσει, εν περιπτώσει, κάτι από πλευρά του Συμβουλίου. δεύτερα, να αποφασίσαμε να υπάρχουν ε, επιδοτήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε ό,τι αφορά τέτοια λειτουργικά και ζητήματα. και στα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το επιθυμεί αυτό. Το Συμβούλιο ενδεχομένως να ήταν ε, πιο ανεκτό, αλλά εφόσον δεν ε, το επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τελική ανάλυση δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ενδεχομένω να πρέπει να αποτεχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ύστερα, στον τομέα των ε, δαπανών για τα έργα για τρίτε χώρε, εδώ έχει έντονε αμφιβολίες το Συμβούλιο. Υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο επισημάνομαι σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κρίσεων. Εδώ και το Συμβούλιο και η Επιτροπή θέλουν να κινηθούν προς το νέο αυτό εργαλείο για τις φυσικές καταστροφές. Εκεί θέλουν να μας ε, στρέψουν. Αλλά πώς να σας το πω, οι τρομοκρατικές επιθέσεις είναι διαφορετικό πράγμα. Σε τρομοκρατικές επιθέσεις θα πρέπει να είμαστε σε θέση και σε θέματα ασφάλειας να έχουμε μια πολύ στενή και ακριβή συνεργασία. Το θέμα της ε, επίλυσης ε, κρίσεων το είδαμε και τη συνεργασία. Το είδαμε και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στο Βέλγιο στι τρομοκρατικέ επιθέσει. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα τουλάχιστον να σε χρηματοδοτήσουμε αυτά που χρειάζονται. Άλλο θέμα. Κυβερνό έγκλημα και κυβερνό ασφάλεια. Εδώ λοιπόν είχαμε βασικά ζητήματα και στον τεχνικό τριμερή διάλογο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούσαμε πολλά σημαντικά επιχειρήματα. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήθελε να ανοίξει τα χαρτιά τη, παρά το γεγονό ότι το συμβούλιο ήταν μάλλον θετικό. Το θέμα λοιπόν της κυβερνοασφάλεια για την ε, ασφάλεια των πολιτών θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε ό,τι αφορά και την χρήση των μέσων του ESF. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό δεν επιλύσαμε τα ζητήματα τα οριζόντια. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει πιο οριζόντιο χαρακτήρα από ότι εμείς. Ε, αλλά εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν μπορώ να αποκλίνω από την ουσία τη εντολής την οποία μου έδωσε η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Σε αυτό το πνεύμα θα διαπραγματευτώ. Εδώ λοιπόν σε ό,τι αφορά τις οριζόντιες διατάξεις είμαστε πολύ περιορισμένοι και ήταν πολύ περιορισμένη και η πρόοδος που πετύχαμε. Δεν πετύχαμε καμία πρόοδο δηλαδή ουσιαστικά. Και η Φιλανδική Προεδρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, οι τρεις συζητητές, όλοι συμμετέχοντες διαπιστώσαμε μια κάποια πρόοδο ότι αφορά τα θέματα διαφάνειας. Αλλά ειλικρινά προχωράμε με ρυθμούς χελώνας. Και γι' αυτό λοιπόν ζητώ από τους συναδέλφους του εξή. Να μου πούν, έχει νόημα να συνεχίσουμε τους τεχνικούς ε, τριμερείς διαλόγους τη στιγμή που δεν υπάρχει πολιτική βούληση και πραγματικά η πρόοδος είναι μηδαμινή. σε ό,τι αφορά λοιπόν τα θέματα των άλλων υπηρεσιών, σε ό,τι αφορά τι θεωρήσει κλπ. Μήπω να αποτανθούμε γραπτά προ το Συμβούλιο και εγώ προσπαθώ να κλείσω και μία συνομιλία με την Προεδρία. Δεν έχει νόημα να προχωράμε με κάποια στοιχεία. Και στο μεταξύ έχω συνηθίσει και αυτού του τρει διαλόγου που λένε: Ωραία, σημείο ένα στην ημερήσια διάταξη. Ε, θέση του Κοινοβουλίου. Τοποθετούμαστε και πολύ ωραία να ακούσουμε και τι απόψει των κρατών μελών. Δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη, τρίτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Τα ίδια συμβαίνουν και απλά επαναλαμβάνουμε αυτά που ήδη έχουμε ακούσει και αυτά που έχουμε ήδη πει στι προηγούμενε προεδρία και ούτω καθεξή. Και πραγματικά αυτό είναι πολύ δυσάρεστο, είναι δυσάρεστο και για τους υπαλλήλους για το λόγο λοιπόν αυτό θα προσπαθήσω να έρθω σε επαφή με την Προεδρία του Συμβουλίου να του ρωτήσω, μα τι φαντάζεστε, πώς θα προχωρήσουμε. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, με αυτά που κάνουμε δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτε. Ε, σε επαναλήψεις. Και σε κανένα σημείο δεν σημειώνεται πρόοδος. Αυτή η λυπηρή αναφορά από πλευρά μου. Δυστυχώς δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. γιατί ούτε το Συμβούλιο είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένο, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να κάνει ένα βήμα προς τα εμάς, άρα είμαστε λίγο σε σκοτεινά είδατα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή η Προεδρία να προχωρήσει και να καταφέρει να πάρει εντολή και να ευχαριστήσω και τους σκιώδες συζητητές. και δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο και να πετύχω το οτιδήποτε με την ομάδα των ε, εισηγητών. Τι να κάνουμε, εσείς μας ε, παρουσιάσετε την κατάσταση και ζητάτε τη γνώμη σα γιατί είστε πολύ πεπειραμένοι. Και μπορεί να μην είναι ιδεώδη η κατάσταση, αλλά μας παρουσιάσετε τις απόψεις σας και την αξιολόγηση που κάνετε και είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη την πλούσια εμπειρία που έχετε για τα θέματα αυτά. Είναι πολύ σημαντικές οι πολιτικές πτυχές αυτού του θέματος. Σε ό,τι αφορά τους και ηγητές, μόνο ο κύριος Ρωμαίο Φράντς από τους Πράσινους ζήτησε το λόγο. Και αν δεν έχουμε άλλους σκιώδεις ηγητές που να ζητούν το λόγο, α, και ο κύριος Κόφοντ επίσης. Πρώτος γύρος με τους σκιώδεις ηγητές. Ο κύριος Ρωμαίο Φράντς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έλαβα γνώση ότι στι χθεσινέ αντιπραγματεύσει σε τεχνικό επίπεδο η πρόταση για την ε, εκπαίδευση κατά του ρατσισμού τη αστυνομία αφαιρέθηκε από το προσαρτήμα και αναφέρεται μόνο σε μια τελογική σκέψη. Συντόμω. Και δεδομένη τη αύξηση του ρατσισμού στην κοινωνία μα, είναι θεωρώ καθήκον μα σε όλα τα επίπεδα, σε πολιτικό επίπεδο και θεσμικό επίπεδο, να ασκήσουμε οποιαδήποτε πίεση έχουμε στη διάθεσή μας για να καταπολεμήσουμε τον ρατσισμό. Αγαπητή Μόνικα, αγαπητή κυρία Χολμάιερ, δεδομένων και των όσων συνέβησαν χθε στην Θουρικία και σε ό,τι αφορά και την επέτειο τη Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου την προηγούμενη εβδομάδα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω τέτοια μέτρα να μην ε, τα αγνοούμε και στην Κροατία που η αστυνομική βία κατά των μεταναστών είναι κάτι καθημερινό πλέον ως φαινόμενο όπου θα ήταν σωστή και κατάλληλη αυτή η εκπαίδευση κατά του ρατσισμού. Θα ήθελα λοιπόν να μπει αυτό και μάλιστα σε εμφανές σημείο στο κείμενο. Μας, Σας ευχαριστώ κύριε Φράντσο. Κύριο Σκόφωτ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας, την κυρία Χολμάιερ, για το έργο της στην έκθεση αυτή. Είναι πραγματικά άρτιο και μπράβο της. Είναι αμφισβήτητο ότι η ασφάλεια των Ευρωπαίων απειλείται και είχαμε πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις ε, σε μεγάλες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, στο δρόμο, σε μεγάλα εμπορικά κέντρα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να βρούμε τις καλύτερες λύσεις για να προσπίσουμε την εσωτερική ασφάλεια και ακόμη και δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών, θα πρέπει να προωθήσουμε κάποιες ε, καλές πρωτοβουλίες, όπως αυτή που προτείνεται εδώ. Σε ό,τι αφορά τις τρίτες χώρες, είναι σαφές ότι εκεί θα πρέπει να καταπολεμηθούν οι βασικές απειλές, από εκεί που πηγάζουν, από τις τρίτες χώρες. Μερικοί θεωρούν ότι θα πρέπει να τιμωρήσουμε αυτές τις χώρες που εξάγουν τα προβλήματά τους στην Ευρώπη. Και είναι σαφές ότι μερικές φορές η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως εργαλείο κατά των κρατών μέλων. Και βλέποντας την κατάσταση μεταξύ 2014 και 2020, δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω την εισηγήτρια και να συμφωνήσω μαζί της. Θα πρέπει επίσης να δούμε την πολιτική των θεωρήσεων και την πολιτική εξωτερικών συνόρων. Εμείς συμμετέχουμε στις δύο πολιτικές. Είναι σαφές όμως ότι ενισχυμένος έλεγχος των εξωτερικών συνόρων και η σωστή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και του συστήματο των θεωρήσεων είναι απολύτως σημαντικά σημεία και γι' αυτό χρειαζόμαστε το Ταμείο εσωτερική Ασφάλειας. Εσείς είστε υπέρ μια ε, εκχώρησης αρμοδιοτήτων. Αυτή είναι πολύ σημαντική αν θέλουμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστούμε κύριε Κόφωτ. Υπόλοιποι συνάδελφοι τώρα, ο κύριος Μπρέιερ. Ευχαριστώ. Μάλλον παρεξήγηση έγινε. Εγώ δεν ζήτησα το λόγο. Πώς habido un malentendido. Α, παρανόηση. Κυρία Χολμάιερ, ή μάλλον όχι, κάποιος άλλος. Θα είμαι μείωπες, δεν βλέπω. Ο κύριο Ρέσλερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η θέσπιση του Ταμείου εσωτερική ασφάλεια είναι αναφυσβήτα προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Εγώ είμαι η συγκητή τη Επιτροπή τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για τον προπολογισμό του 2021 και θα φροντίσω να λάβω υπόψη μου τη θέση μα στον επόμενο προπολογισμό. Έχουμε όλο και περισσότερε απειλέ στην ασφάλεια στο, στο ραγδαίο εξελισσόμενο κόσμο και αυτό ισχύει στην, ε, στο κυβερνοέγκλημα, το ξέπλυμα χρήματος και στις όλο και πιο ε, εκλεπτισμένες μεθόδους που χρησιμοποιεί το οργανωμένο, διεθνές οργανωμένο έγκλημα. Γι' αυτό και η εσωτερική ασφάλεια θα πρέπει να βρεθεί ψηλά στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι η προτεραιότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης, και οι πολιτικοί θύνοντες θα πρέπει να εξασφαλίσουν χρηστή διαχείριση όλων αυτών των ταμείων και των συναφών κονδυλίων. Και θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο στο Συμβούλιο για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Δυστυχώς όμως είναι δεμένα τα χέρια της Κροατικής Προεδρίας στο Συμβούλιο και όλες οι προτάσεις το έχουν την περικοπή των κονδύλιων, κάτι που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Επίσης, ειλικρινά πιστεύουμε και ελπίζουμε η Κροατική Προεδρία να έχει πλήρη εντολή στις διαπραγματεύσεις για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ώστε να καταφέρουμε εγκαίρως ε, να εγκρίνουμε τη θέσπισή του. Ευχαριστώ. Κύριε Χολμάιρ. Να σας ευχαριστήσω αγαπητοί συνάδελφοι καταρχάς για τις τεχνικούς τρεμερείς διαλόγους δεν γίνονται οποιασδήποτε τελειωτικές ε, οριστικές συμφωνίες. Αυτές οι πληροφορίες δεν στέκουν. Όλα αυτά που συζητιούνται ε, στους τρεμερείς τεχνικούς διαλόγους ε, συζητιούνται στη συνέχεια και από τους σκιώδες εισηγητές και στη συνέχεια αποφασίζεται τι θα γίνει. Δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή το οριστικό στην παρούσα φάση. Δεν χρειάζεται λοιπόν να αποσύρουμε και τίποτα. Νομίζω ότι υπάρχει μια πρόταση ωστόσο προς την κατεύθυνση αυτή και θα ήθελα να καταλάβω γιατί και πώς, γιατί δεν το καταλαβαίνω απόλυτα. Θα ήθελα λοιπόν να τα συζητήσουμε, αλλά εγώ δεν έχω λάβει σχετική απάντηση. σε κάποιους τομείς, δυστυχώς, δυστυχώς δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος και όλα προχωρούν με πολύ αργούς ρυθμούς. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις τις οποίες θα τις εξετάσουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναδέλφους και τον για την υποστήριξή του. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε όντω να λάβει η κρατική προεδρία μια πλήρη πραγματική εντολή, γιατί ιδάλω δεν έχει κανένα νόημα να γίνονται αυτές οι τριμερείς ε, τεχνικές συζητήσεις. Χαμογελάμε όλοι, είμαστε όλοι ευγενικοί, αλλά γενικά προκαλούνται έντονα συναισθήματα και αγνακτήση προφανώς και Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει αυτή η κρατική προεδρία να λάβει μια αντιπραγματευτική εντολή με την οποία να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλά λέει ο πρόεδρος. Επομένως η συγκεκριμένη πρόταση ακόμα ισχύει ε, στο ύψιστο ε, επίπεδο δεν έχει ε, απορριφθεί και έτσι να σταματήσουν να γίνονται ξανά και ξανά τα ίδια. Επομένω, εμεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε, τόσο ώστε αυτό που θέλετε να έχει αίσια κατάληξη. Άρα θα τα λέμε σε αυτά που είπατε και θα προσπαθήσουμε να διεκπεριώσουμε τη, τη, την ε, προσπάθειά σα όπω πρέπει. Ευχαριστούμε. Κάτω τούτου. Δεν έχουμε άλλα σημεία στη μεσαία Δεξιού, οπότε πρέπει να σα πω ότι η προσχέση τη συνδρέση είναι 19 Φεβρουαρίου 9 με 12.30 και 3 με 6.30 στις Βρυξέλλες και στις 20 Φεβρουαρίου 9 με 12.30 και 2 με 5,5 στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα στην συνεδρία σας.